So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Συνάδελφοι, καλημέρα σα. Να ξεκινήσω με τι ανακοινώσει. Ε, Εκτό από εστονικά και μαλτέζικα έχουμε όλε τι γλώσσε σήμερα, ούτε κροάτικα δεν έχουμε δυστυχώ. Αλλά σήμερα το απόγευμα και δυστυχώς θα χρειαστεί να αλλάξουμε αίθουσα. Σήμερα το απόγευμα θα τα πούμε στην ε, γνωστή μας ε, ε, αίθουσα. Αλλά την απασχολείται αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Απασχόληση, γιατί είναι μεγάλη η, διάστη, η μεγάλη συνεδρίαση. Να καλωσορίσω ένα νέο μέλο, Κλάου Λάζεν Γένσεν. Καλώ ορίσατε, ο Κλάου Λάζεν Γένσεν. Τον κύριο Γιώργενσον αντικαθιστά ο οποίος μας έγκαταλείψε μέσα Δεκεμβρίου, έγινε υπουργό στην Δανία. Άλλη ανακοίνωση. Τέταρτη ανακοίνωση. Έχουμε ένα εργαλείο στο ίντερνετ ε, όπου μπορούμε να κάνουμε σχετικές αιτήσει. Είναι μια προσπάθεια μέχρι την Παρασκευή 24 ε, Ιανουαρίου. Αν χρειάζεται βοήθεια, αν χρειάζεστε βοήθεια, να απευθυνθείτε είτε στους ε, ε υπαλλήλους της Επιτροπής, είτε σε άλλους συναδέλφους που γνωρίζουν το, το εργαλείο για να το βελτιώσουμε, εν πάση περιπτώσει. Πέμπτη ανακοίνωση. Έχουμε ψηφίσει στην Ολομέλεια την ε, οδηγία για το μέλι το Μάρτιο θα γίνει η τελική ψηφοφορία. Δεν βλέπω ομάδες επισκεπτών ακόμη. Έχουμε και μία ομάδα, μια ομάδα που περιμένουμε τον συνάδελφο Καλ Χάιντς ε, Φλόρενς και τη κυρία Σοφή Οκονή, αλλά δεν έχουν έρθει ακόμα. Να συνεχίσουμε λοιπόν στο 8ο σημείο της ανακοινώσεων. Το εργαστήρια για την υγεία του, της κυρίας Βίλμοντ και του κυρίου Πέτερλε θα λάβει χώρα την Τρίτη από τις 12.30 στο PH 7005. Και συνεχίζω σήμερα. Πρέπει να αντικαταστήσουμε έναν αντιπρόεδρο σας ανακοίνωσα πριν από λίγο, ο κύριος Γιώργενσεν ε, έφυγε από την Επιτροπή μας και από το Κοινοβούλιο. Και τώρα λοιπόν θα πρέπει να αντικαταθήσουμε την ε, θέση του. Προτάσεις λοιπόν, υποψηφιότητες. Η Λίντα. Λυπάμαι που έφυγε ο Γιώργενς, ένα εξαιρετικό μέλος και εξαιρετικός ε, αντιπρόεδρος και έγινε τώρα υπουργός να καλωσορίσω τον Λάρσεν Γένσεν και θα ήθελα να τον προτείνω για αντιπρόεδρο. He has long background in European affairs. Έχει πείρα στα ευρωπαϊκά θέματα. Ήταν πρόεδρος ε, της Επιτροπής για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις στο Folketing. Και είμαι βέβαια ότι θα γίνει ένας εξαιρετικός αντιπρόεδρος για το λίγο καιρό που έχουμε ακόμα. Σας ευχαριστώ για την υποψηφιότητα. Να ρωτήσω λοιπόν και τον υποψήφιο, τον Κλάους Κλάρσεν Γένσεν, κατά πόσον προτίθεται να αποδεχτεί. Αποδέχομαι, απαντάει ο κύριος Λάρσεν Γένσεν. Μάλιστα λοιπόν, διαβοής λοιπόν. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας και χαίρομαι που πλέον είμαστε πλήρεις. Και μπορούμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Το 4 της της διαταξής. Gut, weiter geht's. Und zwar das Protokoll vom 14. November 2013. Τα πρακτικά τη 14 η Νοεμβρίου 2013 εγκρίνονται, εάν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσει, Θεωρώ ότι εγκρίνονται και καλωσορίζω λοιπόν τον Υπουργό. So, ich begrüße ganz herzlich den griechischen. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον ε, Έλληνα Υπουργό Υγεία, ε, τον κύριο Γεωργιάδη. Έχουμε διάφορα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Βλέπω και τη συνάδελφο Ροντ Μπέρεν που είναι εδώ για, τα, ε, για τον ιατρικό εξοπλισμένο, για τον κύριο Πατερλίζα Βλέπω επίσης που είναι υπεύθυνο για τα, τον εξοπλισμό διαγνωστική. Έχουμε την εξή διαδικασία την οποία και ακολουθούμε. Σας δίνουμε το λόγο για την παρουσίασή σας και στη συνέχεια ξεκινάμε με τους συντονιστές από τις ομάδες για ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων. Θα έχετε στη συνέχεια τη δυνατότητα να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Να μην σας καθυστερήσω άλλο. Θα ήθελα να σας δώσω πάρα λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους βουλευτές που είναι εδώ σήμερα μαζί μου. Κυρίε και κύριοι, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να είμαι σήμερα εδώ με την ευκαιρία της ανάλυσης Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απευθύνομαι σε εσά ως βασικούς συντελεστές του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος αλλά και εκφραστές της βούλησης των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πέμπτη φορά μετά την ένταξή σε ευρωπαϊκές κοινότητες το 1981 σε μια μεταβατική περίοδο και ένα πολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σημαντικές προκλήσεις για την Ελλάδα αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη δοκιμάστηκε διάρκεια των τελευταίων ετών, το ίδιο και οι πολίτες της, ενώ η εφαρμογή πολιτικών αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχία επηρέασε την κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερα στις χώρες που αντιμετώπισαν την κρίση άμεσα, όπως η χώρα μου, η οποία δοκιμάστηκε ίσως όσο δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωση. Έχουμε όμως ήδη τα πρώτα σημάδια ότι η κρίση αυτή αρχίζει να ξεπερνιέται. Η Ελλάδα, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ύφεση, εξέρχεται από την οικονομική κρίση και κατευθύνεται πλέον προς την ανάκαμψη. Ωστόσο η κρίση δεν έχει τελειώσει. Η ανεργία συνεχίζει να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε αρκετά κράτη-μέλη πλήττοντα ιδιαίτερα του νέους, στη δική μου χώρα πάρα πολύ, με την ανάπτυξη να είναι το ζητούμενο. Και όλα τα παραπάνω, μόνο τέσσερι μήνε πριν τι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίε συνιστούν έναν πρόστο παράγοντα που ορίζει το πλαίσιο τη Προεδρία μα. Το μεγάλο διακύβευμα είναι η επιβεβαίωση της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καρδιά και στον νου των πολιτών της. Με γνώμονα τα ανωτέρω και προκειμένου να απαντήσουμε αποτελεσματικά στην κρίση και στον αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό. Τις προτεραιότητες προεδρίας μας παγορεύουν οι ανάγκες των πολιτών της Ένωσης και συνοψίζονται στα ακόλουθα, θέματα, τέσσερα θέματα. Πρώτον, στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεύτερον, στην εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με τη στήριξη του κοινού μας νομίσματος και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τρίτον, στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης της μετανάστευσης και τέρτον στις θαλάσσιες πολιτικές στις οποίες φιλοδοξούμε να δώσουμε μια νέα πνοή. Αντίστοιχα θα κινηθούν και οι προτεραιότητες μας στον τομέα της υγείας. Αναγνωρίζοντας ότι η καλή υγεία αποτελεί προϋπόθεση για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, θα εργαστούμε προκειμένου να υπάρξει πρόοδος με στόχο την ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου και την προώθηση πρωτοβουλειών και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για περισσότερα αποδοτικά συστήματα υγείας και καλύτερη υγεία. Στο νομοθετικό πεδίο θα ήθελα πρωτίστως να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής σε μια εξόχως σημαντική νομοθετική πρόταση, στην πρόταση οδηγίας για τα προϊόντα καπνού και ευελπιστώ το ίδιο θετική θα είναι και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ίδιο και για την πρόταση για τι κλινικέ δοκιμέ, την οποία θεωρούμε σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη τη κλινική έρευνα. Κεντρική θέση στι εργασίε επομένη περίοδου θα έχουν οι προτάσει για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Πολύ σημαντικέ προτάσει, οι οποίε θα βελτιώσουν την ασφάλεια των ασθενών μέσω τη ενίσχυση των διαδικασιών προεγκριτικού ελέγχου και μετεγκριτική επιτήρηση αγορά. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ χρηστών, επαγγελματιών υγείας και οικονομικών φορέων είναι υψής της σημασία για την ευρεία χρήση, την απρόσκοπτη κυκλοφορία και την ενθάρρυνση της καινοτομίας. Τα επιτεύγματα της ιατρικής τεχνολογίας μπορούν να δώσουν όθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με παράλληλη μείωση του κόστους και ενίσχυση αποδοτικότητας της υγειονομικής περίθαλψης. Θα συνεχίσουμε το έργο των προηγούμενων Προεδριών και δεσμευόμαστε να επιδιώξουμε να υπάρξει σημαντική πρόοδο και αν είναι δυνατόν και συμφωνία. Για το σκοπό αυτό έχουμε καταρτήσει ένα πρόγραμμα εντατική εργασία για το διάστημα των επόμενων μηνών. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση σε επίπεδο ομάδο εργασία Συμβουλίου με θετικά πρώτα αποτελέσματα. Στην πρόταση για τέλη φαρμακοεπαγρύπνηση, η οποία αποβλέπει να παράσουν Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων τα απαραίτητα μέσα για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που προβλέπει η νέα νομοθεσία, προσδοκούμε στην επίτευξη συμφωνία εντό του επομένου μηνό, ώστε η νέα νομοθεσία να ισχύσει από τον Ιούλιο. Σήμερα, σε στο Κορεπέρ, το αίτημά μα για παραχώρηση εντολή έναρξη του τριμερού διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Ευελπιστώ ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και ο προγραμματισμένος αυριανός πρώτος τρίλογος θα είναι επιτυχής. Τέλος, θα επιδιώξουμε πρόοδο στην οδηγία για τη διαφάνεια, η οποία αποβλέπει στην εξασφάλιση διαφάνειας, στην τιμολόγηση και αποζημίωση, στην βελτίωση της πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα και στη διευκόλυνση θέση στην αγορά των γενοσύμων φαρμάκων, καθώς και στην ενθάρρυνση της έρευνας και ανάπτυξης του φαρμακευτικού τομέα. Στο μη νομοθετικό πεδίο τώρα, οι προτεραιότητες μας θα εστιάσουν στους ακόλουθους τέσσερι αρχές. Πρώτον, οικονομική κρίση και υγειονομική περίθαλψη. Έχοντας επίγνωση της οικονομικής κατάστασης και των επιπτώσεων στην υγειονομική περίθαλψη και στα συστήματα υγείας, έχουμε θέσει ως πρώτη γραμμή προτεραιότητας το θέμα της αποδοτικότητας και βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, η δική μας χώρα έχει μια μεγάλη εμπειρία αυτό το θέμα αυτά τα τελευταία τρία χρόνια για προφανείς λόγους. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο των συζητήσεών μα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Υγεία στα τέλη Απριλίου στην Αθήνα. Θα εστιάσουμε κυρίω στο πώ ανταποκρίθηκαν τα συστήματα υγεία σε περίοδο οικονομική στενότητα σε επίπεδο προπολογισμών, μεταρρυθμίσεων και υγειονομικών αποτελεσμάτων ω προ την πρόσβαση, την ποιότητα των υπηρεσιών και την ανταποκρισιμότητα των πολιτών στην Ελλάδα υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και έχουμε ήδη θετικά αποτελέσματα σε τομείς όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ενώ σημειώσουμε σημαντική πρόοδο στον τομέα του εξορθολογισμού των δαπανών και εξυγχρονισμού του νοσοκομιακού τομέα. Θα ήθελα σε αυτόν τον τομέα ιδιαίτερα να σημειώσω την πολύ θετική συμβολή της Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτών των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση την αναδιάρθρωση τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Ενώ έμφαση δίνουμε στην υγειονομική κάλυψη των περισσότερων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Μάλιστα αυτή την Παρασκευή εισάγουμε στο Εθνικό μα Κοινοβούλιο το σχετικό νόμο που έχουμε δημιουργήσει και με τι συμβουλέ του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγεία. Αντίστοιχε μεταρρυθμίσει βρίσκονται σε εξέλιξη και στα άλλα κράτη-μέλη. Έχει γίνει πολλή δουλειά και έχουμε επιτυχημένα παραδείγματα. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει αξιολόγηση διδαγμάτων προσδιορισμός των πρακτικών και εν τέλει ανάδειξη των βασικών σημείων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το ιδανικό πακέτο μέτρων πολιτικής αντιμετώπισης κρίσης και κατάρτισης του μοντέλου ανάκαμψης. Στη βάση των ανωτέρων συζητήσεων και του έργου των προηγουμένων Προεδριών θα προωθήσουμε συμπεράσματα Συμβουλίου. Δεύτερον, μετανάστευση και δημόσια υγεία. Στόχος ελληνικής Προεδρίας είναι να θέσει το θέμα της μετανάστευσης και των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία στο επίκεντρο των συζητήσεων. Θεωρούμε ότι απαιτείται συνολική διαχείριση του προβλήματος αυτού, που ναι μεν ενθύγει περισσότερο κάποιες από τις χώρες που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της Ένωσης, αφορά ωστόσο όλους, γιατί οι ασθένειες δεν γνωρίζουν σύνορα. Οι αρχές που πρέπει να διέπουν την προσέγγισή μας είναι η αλληλεγγύη και η αναλογικότητα στην κατανομή των βαρών στη φροντίδα υγείας ταλαιπωρημένων ανθρώπων θα επιδιώξουμε μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κάλυψη των αναγκών υγεία των μεταναστών, τι επιπτώσει στα συστήματα υγεία και του κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Και κυρίω την προβολή των θετικών πτυχών μια ενισχυμένη συνεργασία στην αντιμετώπιση μια κοινή πρόκληση. Τρίτον, η διατροφή και η φυσική άσκηση. Δύο από του σημαντικού παράγοντε μπορούν να καθορίζουν το συνολικό επίπεδο υγεία. Στόχο μα, η ανάδειξη τη υγιεινή διατροφή σε συνδυασμό με τη φυσική άσκηση ως επιλογές υγιούς συμπεριφοράς τρόπου ζωής καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της ζωής από την παιδική ηλικία μέχρι την τρίτη ηλικία στο ευρύτερο πλαίσιο της μάχης κατά της επιδημίας των χρονίων νοσημάτων. Σκοπεύουμε να διοργανώσουμε υπουργική διάσκεψη στις 25-26 Φεβρουαρίου και να υποβάλουμε συμπεράματα Συμβουλίου. Και τέταρτον, η ηλεκτρονική υγεία. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και σε λύσεις ηλεκτρονικής υγείας που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας. Θα φιλοξενήσουμε έκθεση για την ηλεκτρονική υγεία 2014, αποσκοπώντας την όθηση της ψηφιακής ατζέντα και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων λύσεων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναμόρφωση των συστημάτων υγείας, στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης, στην ενδυνάμωση των ασθενών, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Βλέπουμε ότι τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες μήνες θα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Εμείς βρισκόμαστε σε μία φάση όπου θα συνεδριάσουμε μέχρι το Πάσχα. Σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα λοιπόν έχουμε διοργανώσει και τριμερείς διαλόγους προκειμένου να ε, προχωρήσουμε τα ζητήματα τα οποία ήδη έχουμε ξεκινήσει, τα οποία είναι κρεμία ακόμα, προκειμένου να τα κλείσουμε στο βαθμό του δυνατού. Και λοιπόν σας ευχόμαστε και μας ευχόμαστε καλό κουράγιο. Να ξεκινήσουμε με τον γύρο των συντονιστών, ο κύριος Πέτερ Λίζε και η κυρία Ντάγμαρ Ροντμπέρεντ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την δουλειά σα, ε, για το έργο σα. Είχαμε την ευκαιρία ε, να μιλήσουμε και νομίζω ότι ξεκινάτε πολύ δυναμικά την Προεδρία. Δύο θέματα ήθελα να αναφέρω. Καταρχά, είπατε ότι η κρίση σταδιακά ξεπερνιέται. Νομίζω ότι υπάρχουν και αριθματικά στοιχεία, γεγονότα, περιστατικά ε, που το καταδεικνύουν να Έχει πλεόνασμα και μάλιστα ρευστικό πλεόνασμα η Ελλάδα. Πιο πολλά έσοδα από δαπάνε σε Μία κατάσταση την οποία ούτε καν ονειρεύεται η Αμερική για παράδειγμα. Και Όλοι όσοι προβλέπαν ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα και ότι θα πρέπει να βγει η Ελλάδα από το ευρώ, διαψεύστηκαν. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την θυσίες σας. Ξέρουμε τις θυσίες που έγιναν, αλλά στέφθηκαν με επιτυχία και αυτό επιβραβεύει και την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Στο θέμα των ε, Τη υγεία, σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Πριν από κάποια χρόνια λάβαμε την πληροφορία ότι για παράδειγμα στην Ελλάδα ε, χρησιμοποιούνται πάρα πολύ λίγα γενώσιμα φάρμακα και ότι χρησιμοποιούνται τα πολύ ακριβά ε, πρωτότυπα. Ήταν δύσκολη λοιπόν η κατάσταση. Πώς το αντιμετωπίσατε λοιπόν και σε ποια φάση βρίσκεστε σε, αυτό το θέμα. Δεύτερο ζήτημα σε ό,τι αφορά ε, τα ε, προϊόντα και τον εξοπλισμό μικροδιαγνωστικών. Ε, στις, ε, γίνεται ένα τριμερής διάλογο θα θέλαμε να τον ολοκληρώσουμε πριν από τι ευρωεκλογέ και για τον κλάδο και για τις ε, ασθενεί. Αν δεν περάσει, αν δεν τα καταφέρουμε, θα σα καλούσα να συμπεριλάβετε όσο πιο πολλά γίνεται από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και σε ό,τι αφορά και τα συμπεράσματα της κυρίας Ροτ Μπέιρεντ, ε, στη δική μου έκθεση το θέμα της ε, ενήμερης ε, συνένεσης σε ό,τι αφορά τα τεστ DNA. Το συζητήσαμε. Μέχρι και στην Αμερική είναι πάρα πολύ έντονη η κριτική που ακούγεται κατά πόσον πρέπει και να επιτρέπεται η διαγνωστική αυτή μέσω διαδικτύου χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη προετοιμασία και υπάρχει ανησυχία εδώ στο Κοινοβούλιο ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βλάψει πιο πολύ τον άνθρωπο αν δεν ρυθμιστεί σωστά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ροτπέραντ, σας ευχαριστώ Ματίας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γεωργιάδη, τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου πλέον. Θαυμάζω και εγώ από πλευράς μου για το τι καταφέρατε να κάνετε στην χώρα σας, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, έναν πάρα πολύ δύσκολο τομέα. Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει και ο τομέας της υγείας είναι ένας τομέας ο οποίος θίγει τους ιδιαιτέρως ε, εύθραστους αν θέλετε τα ιδιαίτερως εύθραστα τμήματα του πληθυσμού, οι οποίοι θίγονται περισσότερο από τους υπόλοιπους πολίτες και το να καταρρεύσει, να καταρρεύσει ο τομέας της υγείας θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κάνατε και χάρη στις δικές σας προσπάθειες και στις προσπάθειες της κυβέρνησής σας υπάρχει δρόμος ακόμα Είπατε ότι η καλή υγεία είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία της κοινωνίας. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και σε άλλες χώρες. Και ε, θα πρέπει να βάλουμε στην επόμενη συνθήκη ότι θα πρέπει να έχουμε αν όχι ίδιες τουλάχιστον συγκρίσιμες συνθήκες στήριξης για αυτούς που έχουν ιατρικές ανάγκες. Και η κοινωνία, η ελληνική γενικότερα Νομίζω ότι ε, ξέρω ότι θα ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση για τη χώρα σας αν πράγματι δεν χρειαζόταν να επιστρέψουν τις πιστώσεις τις οποίες είχαν πάρει όλα αυτά τα χρόνια σε χώρες όπως η δική μου και να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν. Επανέρχομαι όμως στο παρόν. Όπως έχουμε ήδη δίμερο συζητήσει θα πρέπει να αναφερθώ στα θέματα ε, του ιατρικού εξοπλισμού. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Γνωρίζω ότι κάποιες χώρες ε, καθυστερούν. Οι χώρες οι οποίες είναι πολύ διστακτικές είναι πάρα πολύ γρήγορες στον τομέα της φαρμακοεπαγρύπνησης ε, εγώ είμαι πάρα πολύ καχύποπτη, δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο, απλά βλέπουν ναι, τι επιστροφές οικονομικές ε, επανέρχονται στις χώρες λόγω ακριβώς της εφαρμογής της φαρμακοεπαγρύπνησης. Μια μη ε, σωστή πολιτική παρατήρηση αυτό που έκανα. Υπάρχει κάποιος δισταγμός από πλευράς των κρατών μελών όπως αυτός ε, που έδειξαν λοιπόν ε, τους τελευταία, τα τελευταία χρόνια για τους ε, διαγνωστικούς και ιατρικούς εξοπλισμούς και τόσο όσο καθυστερούσαν τότε τόσο βιάζονται τώρα οι ίδιες αυτές χώρες για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και αυτό με ενοχλεί. Θα πρέπει να σταματήσουν οι μεταφορές χρημάτων από την φαρμακοεπαγρύπνηση εφόσον κολλησιεργούν σε άλλους τομείς. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι οι χώρες καθυστερούν, πολλές χώρες μέλη καθυστερούν και απαιτείται να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πιέσει. Η Λιθουανική Προεδρία ήταν φιλόδοξη αλλά πολύ ευγενική και δεν το πέτυχε. Εσείς ελπίζω να είσαστε λιγότερο ευγενικοί. Αυτό δεν θα κάνει τον κόσμο να μη σας αγαπήσει. Και αν θέλουμε να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας το, σε, σε τι θα καταλήξουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι χωρίς καμία καθυστέρηση. Άκουσα ότι εσείς θα είσαστε έτοιμοι στα μέσα Φεβρουαρίου, το αργότερο. Και θα πρέπει επίσης και ε, το δεύτερο κεφάλαιο, το τρίτο κεφάλαιο όπως επίσης και το 5 που είναι το σύστημα έγκρισης. Ε, σε όλα αυτά θα πρέπει να βρούμε μία συμφωνία και θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Λίζα αναφέρθηκε στο θέμα των αλλαγών. Πρόσφατα μια δικαστική απόφαση επιβεβαίωσε την προηγούμενη ε, απόφαση που είχε ληφθεί στην Γερμανία σχετικά με τους μηχανισμούς πιστοποίησης, τους ειδικού μηχανισμούς πιστοποίησης και τις αποζημιώσεις. Αυτά για τους μηχανισμούς κοινοποίησης λοιπόν. Θα ήθελα τώρα κύριε Προεδρεύοντα να μάθω αν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε ένα τριμερή διάλογο. Ξέρετε ότι μπορούμε και εμείς ε, να ψηφίσουμε αρκετά σύντομα στην Ολομέλεια. Αλλά τι εγγυήσει θα έχουμε ότι η υπόλοιπη νομοθετική εργασία με την οποία δεν έχουμε ακόμα ασχοληθεί ε, δεν θα την αγνοήσετε και θα ασχοληθείτε μαζί της το ταχύτερο δυνατόν. Ξέρω ότι όλα αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες και για την Προεδρία, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει μια δήλωση από πλευράς της Προεδρίας ως ειλικρινούς ενδιαμέσου σε όλα αυτά τα θέματα για να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε, αλλά ό,τι κνάνε να γίνει πρέπει να γίνει γρήγορα. Σας ευχαριστώ. Η συνάδελφό πάντα είναι, η συνάδελφό πάντα είναι τόσο ευγενική. Η Ρεμπέκα Τάιλερ. Uh, thank you, Chair. Um, Ευχαριστώ. Προβληματική κατανάλωση αλκοόλ και εξάρτηση από το αλκοόλ σε με 60 χρόνιες νόσους, καρδιαγγικές, διαβήτη, ε, ασθένειες ε, ε, του ύπατος στην Ελλάδα. Εκτιμάται ότι 1,3% και 2,2% των αντρών έχουν μια τέτοια εξάρτηση και το Συμβούλιο επανειλημμένα έχει τονίσει την ανάγκη να μειωθεί κατανάλωση του αλκοόλ. Προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ολοκληρώθει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. πώ θα επεξεργαστείτε σε αυτό το σχέδιο και πώ θα επιτύχετε την απαιτούμενη έγκριση από πλευρά του Συμβουλίου για την εθνική αρμοδιότητα γνωστών. Σα ευχαριστώ από του πράσινου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Εύχομαι να πετύχετε ε, σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση όπως είναι τα θέμα της υγείας με δεδομένο και ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Δηλαδή έχετε να διαχειριστείτε θέματα ευρωπαϊκά την ίδια στιγμή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα στην Ελλάδα ε, όπως το γεγονός ότι υπάρχουν 3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι σήμερα, το 30% του πληθυσμού δεν έχει ασφάλιση για να μπορεί να έχει πρόσβαση στα συστήματα υγείας, που σημαίνει ότι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο άτομα δεν έχουν καμία πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σήμερα και είναι άτομα τα οποία πλήρωναν κανονικά τι ασφαλιστικέ του εισφορέ για πολλά χρόνια. Έχουμε αύξηση 30% εισαγωγών σε νοσοκομεία, Έχουμε τρία, πέντε νοσοκομεία τα οποία έκλεισαν πρόσφατα. Πολλά νησιά και περιοχέ δεν έχουν γιατρού σήμερα και υπάρχουν προβλήματα στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση και μεγάλο, μεγάλο ποσοστό παιδιών εμβολιάζονται σε ιδιώτε ή δεν εμβολιάζονται καθόλου. Πρέπει λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική προεδρία να πετύχει και να λύσει προβλήματα στη χώρα μα, αλλά κυρίω να πετύχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχουμε θέσει και εμεί οι πράσινοι εδώ στην Επιτροπή ΕΝΒΗ είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αισθημάτων υγείας σε περίοδο κρίσης και των μεταρρυθμίσεων που ασκούνται σε διάφορα αισθήματα υγείας. Είναι μια ιστορία που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα ή την Πορτογαλία ή την Ισπανία, αφορά και άλλες χώρες που έζησαν παλιότερα την κρίση, όπως είναι η Φιλανδία, η Γερμανία κλπ. Άρα πρέπει να αξιολογήσουμε τις μεταρρυθμίσεις και αυτό με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Δεν ξέρω αν έχετε, αν έχετε προγραμματίσει ε, μια ειδική σύνδεση που δεν θα είναι μόνο μεταξύ των Υπουργών, του Συμβούλιο, αλλά και με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων από όλη την Ευρώπη. Έχουν γίνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάρα πολλέ τέτοιε εκδηλώσει και οι γιατροί του κόσμου και πολλοί άλλοι φορεί έχουν παρουσιάσει συγκλονιστικά στοιχεία και δεν αφορά η κρίση μόνο την Ελλάδα. Ε, μια ιδιαίτερη παράμετρος αυτού είναι επιπτώσεις στην υγεία σε βάλλοντες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή έχει χειροτερέψει η κατάσταση και έχω δει στοιχεία όχι μόνο για τι χώρε κρίση, αλλά και για τη Γαλλία ή για την, ε, το Βέλγιο κλπ. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια πλήρη εικόνα πανευρωπαϊκή για τα θέματα. Το δεύτερο νομίζω που είναι σημαντικό και αφορά και την Επιτροπή μα είναι τα θέματα τη κλιματική αλλαγή και των επιπτώσεων στην υγεία από την κλιματική αλλαγή και στη χώρα μας έχουμε παραδείγματα όπως ο, ο, ο πυρετός του Νείλου και διάφορα άλλα που ήταν παλιότερα σε άλλες κλιματικές ζώνες. Τώρα έχουν έρθει στη δικιά μας κλιματική ζώνη παρόμοιες ασθένειες, στο εύκρατο κλίμα. Και εν ώψη του Μαΐου του 2015 που υπάρχει η Μεγάλη Σύνοδο στο Παρίσι, ελπίζω ότι η Προεδρία θα οργανώσει ένα μεγάλο ε, γεγονός που θα αφορά την υγεία και την κλιματική αλλαγή. Και το τρίτο θέμα αφορά τη μετανάστευση, όπως είπατε κι εσείς. Είναι σωστό το θέμα της αλληλεγγύης, ε, να κυριαρχήσει πολιτικέ πολιτικές για τη μετανάστευση. Υπάρχουν όμως διάφοροι μύθοι ότι, πολλές, ότι Κοίτα, χρησιμοποιούν, βέβαια αυτού του μύθου χρησιμοποιούν πολλέ φορέ ακροδεξιέ οργανώσει ότι οι μετανάστε κουβαλούν πάρα πολλέ ασθένειε. Έχετε εσεί παρόμοια στοιχεία, γιατί εγώ τουλάχιστον που το έχω ε, διερευνήσει, δεν ισχύει αυτό. Απλώς είναι ένας μύθος που κυκλοφορεί μεταξύ των ακροδεξιών οργανώσεων για να πούν ότι αυτοί μας φέρουν και ασθένειες. Από την άλλη μεριά βέβαια πολλές φορές οι μετανάστες μένουν εκτός των συστημάτων υγείας, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα θέματα. Τώρα τελευταία η Ελλάδα έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τέτοιου πόρου. Ε, για παράδειγμα, όταν μπαίνουν μετανάστε σε μια χώρα, να, γίνεται, ε, να υπάρχει συνεργασία με τα νοσοκομεία για να υπάρχει ας πούμε, μια πλήρη εικόνα τη υγεία του και τι βοήθεια χρειάζονται κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η Μαρίνα Γιανακουδάκη από το ECR. Um, ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια προς την Ελληνική Προεδρία. Προβλέπω ότι θα είναι μια πολύ επιτυχής Προεδρία και γνωρίζω ότι είσαστε πολύ ικανός για να το πετύχετε αυτό τους επόμενους έξι μήνες να ξεκαθαρίσω για τους συναδέλφους μου. Είπαν ότι οι Έλληνες υπέφεραν. Οι Έλληνες δεν υπέφεραν, υποφέρουν, συνεχίζουν να υποφέρουν σήμερα. Οι δείκτες οικονομικοί μπορεί να βελτιώνονται, αλλά ο λαός εξακολουθεί να υποφέρει, πολλούν ό,τι μπορούν τα έπιπλά για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Λοιπόν, η κυβέρνηση κάνει προσπάθεια σημαντική, αλλά ο λαός υποφέρει ακόμα. Εγώ ε, ευχαριστώ την Ελλάδα και για τους γιατρούς που έρχονται στην Αγγλία για να ασκήσουν το επάγγελμα. Έχουν πολύ ψηλό επίπεδο και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια διαρροή εγκεφάλων από την Ελλάδα στον τομέα αυτό και στον τομέα αυτό και αυτό είναι λυπηρό για την Ελλάδα. Λόγω των προβλημάτων λοιπόν που αντιμετωπίσατε τα τελευταία τρία χρόνια, πώς θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη εμπειρία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, γιατί υπάρχουν πολλές χώρες μέλη με οικονομικά θέματα, με προβλήματα. Πώς ε, τα έχετε καταφέρει μέχρι τώρα ε, με τις μεταρρυθμίσεις που κάνατε λόγω της λιτότητας ε, στη χώρα σας. Αναφερθήκατε και στο θέμα της μετανάστευσης και των συνεπειών της στο θέμα της υγείας. Ε, γνωρίζω ότι στην Ελλάδα τα σύνορα δεν είναι πάντα ασφαλή και δεν είναι, υπάρχει εν πάση περιπτώσει μια κάποια παράνομη μετανάστευση. Σε ποιο βαθμό επηρεάζει την υγεία, την δημόσια υγεία. Ξέρω ότι σε κάποιες περιοχές είχαν υπάρξει από μετανάστες αυξήσεις των ποσοστών φυματίωσης, ενώ στο παρελθόν είχαν κρυζωθεί όλα αυτά. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι προκλήσεις έχετε αντιμετωπίσει και στον τομέα της μετανάστευσης και πώς εσείς τα έχετε καταφέρει μέχρι τώρα. Κύριε Υπουργέ, η αντιλαϊκή πολιτική που περιγράψατε προωθείται διαχρονικά και ενιαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις ε, προηγούμενες προεδρίες, από όλες τις κυβερνήσεις, σε όλα τα κράτη-μέλη της, πριν την εκδήλωση της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και επιταχύνεται σήμερα παντού, ανεξάρτητα αν οι χώρες αυτές είναι υπό επιτήρηση, ανεξάρτητα αν υπάρχουν μνημόνια, ανεξάρτητα το ύψος των δημόσιων ελλημάτων. Γιατί όλα αυτά. Γιατί αυτό απαιτεί η καπιταλιστική ανάπτυξη που στηρίζεται στη δράση των επιχειρηματικών ομίλων, στη διείσδυση σε αυτή την περίοδο, ακόμα παραπέρα των μονοπωλίων, σε αυτό το χρυσοφόρο τομέα για, τα για το κεφάλαιο, όπως είναι η υγεία για να αντιληφθούν οι συνομιλητές μας την κατάσταση που περνάει ο, λαό, ελληνικός λαός, θέλω να επισημάνω επιγραμματικά ορισμένα στοιχεία. Η αντιλαϊκή πολιτική αυτή αποτυπώνεται και στον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό για το 2014 με δραματικές μειώσεις δαπανών στο Υπουργείο Υγείας κατά 19,7% σε σχέση με το 2013 με τη μείωση της χρηματοδότησης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κατά 30%, των δημοσίων νοσοκομείων κατά 32% και της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 15%. Αν κάποιος συνυπολογίσει τις συνολικές δαπάνες τόσο σε ό,τι αφορά το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, της συντάξης και, και στις παροχές υγείας και πρόνοιας, το ποσό ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο 850 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και όλες ότι μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό που θα υποβαθμίσει ραγδαία πέρα από οποιοδήποτε ενέργειες γίνουν την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Σε αυτή την πολιτική οφείλεται πρώτο η υπονόμευση και πρόληψη φορά της υγείας των εργαζομένων από την επιδίνωση των συνθηκών δουλειάς αλλά και κατοικίας. Δεύτερο, μεγάλο ζήτημα απασχολεί είναι το τμήμα των ενός εκατομμυρίων χιλιάδων ανέργων που καθώς και άλλων εκατοντάδων χιλιάδων που έχουν βγει εκτός της δημόσιας ασφαλιστικής κάλυψης η υποχρηματοδότηση των κρατικών νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, των υγειονομικών μονάδων του ΕΟΠΗ και των ασφαλιστικών ταμείων είναι γεγονός. Σημαντική, σημαντικές επιπτώσεις υπάρχουν στις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, η αντεκατάσταση ενός μέρους του, μόνιμου, του μόνιμου προσωπικού με εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, ιδιωτικών συνεργείων και της κοινωνικής εργασίας επιδεινώνουν ακόμα παραπέρα τις συνθήκες δουλειάς αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Την τριετία που μας πέρασε αυξήθηκε η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις δαπάνες για τη φαρμακευτική περίθαψη από το 9% στο 27%. Η εξοικονόμηση ποσών από το κράτος με τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα γίνεται με τη μείωση ενός ελάχιστου μέρους από την υπερκερδοφορία της εχώριας και πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας και από την αύξηση των πληρωμών από τους ασθενείς με το σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων που έχουν προηγηθεί από τις κυβερνήσεις. Τέλος, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι το εξής. Η ίδια αντιλαϊκή πολιτική αποτυπώνεται και στο σχέδιο της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οι προτάσεις των επιστημονικών επιτροπών για διατήρηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ως ασφαλιστικού φορέα, είτε αγοραστή και παραγωγού πολιτή υπηρεσιών υγείας, είτε μόνο αγοραστή υπηρεσιών, όπως τελικά αποφάσισε η κυβέρνηση, αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος αυτής της αντιλαϊκής, αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν ήρθαμε εδώ μόνο να επισημάνουμε σε ό,τι αφορά τις σημαντικές σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τα αντιλαϊκά μέτρα στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας. Αλλά να συνεχίσουμε και να, να διατυπώσουμε ότι διεκδικούμε την ανάπτυξη ενιαίου αποκλειστικά κρατικού και απολύτως δωρεά δημόσιου συστήματος ε, παροχής φροντίδα, πρωτοβα, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με βασικό προσανατολισμό την πρόληψη και με την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να πάρθουν μέτρα. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε για την ε, ε πρώτη αυτή ομιλία εδώ στην Επιτροπή μας. Έχουμε και διερμηνείς, έχουμε και μικρόφωνα. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο ήσυχα και ήρεμα. Ολοκληρώσαμε έτσι λοιπόν ε, τον πρώτο γύρο των ε, ερωτήσεων. Να παρακαλέσω τον Υπουργό να απαντήσει λοιπόν στις ερωτήσεις αυτές και μετά θα περάσουμε κατευθείαν στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων, γιατί έχουμε πολλούς συναδέλφους ακόμα στον κατάλογο. Έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο μπορώ πιο γρήγορα σε όλες τις ερωτήσεις και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους διάστημα τον χρόνο για να μου κάνουν ερωτήσεις. Ε, ξεκινάμε τον κύριο Λίσε. Ε, η κρίση ξεπερνιέται πράγματι και η Ελλάδα είναι, έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια πράγματα που και εμένα με ρωτούσατε αν θα τα καταφέρναμε, δεν θα πίστευα θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε τόσο γρήγορα. Όμως πράγματι πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό έχει γίνει με τρομερές θυσίες των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει να ξέρετε όλοι ότι στην Ελλάδα χάσαμε τα τελευταία τρία χρόνια κατά μέσο όρο το 30% του εισοδήματό μα όλοι οι Έλληνε πολίτε. Και αυτό εύκολα λέγεται σε ένα συμβούλιο, αλλά όταν μια κοινωνία το βιώνει είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει λοιπόν να σα πω ότι δεν έγινε αυτή η αλλαγή τη χώρα χωρί πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και σίγουρα και το αναγνωρίζουμε και χωρί βοήθεια από την Ευρώπη. Γιατί η Ελλάδα έγινε το σύμβολο τη κρίση τη Ευρωπαϊκή Κρίση Χρέου, αλλά η Ελλάδα θα γίνει και μπορεί να γίνει και το σύμβολο τη αλλαγή σελίδα και τη νέα πορεία Ευρωπαϊκή Ένωση προ ένα καλύτερο αύριο. Και το πιστεύουμε ακράδαντα αυτό. Τώρα πάω λίγο στο, στα συγκεκριμένα που μου θέσατε. Ε, στα γενώσμα η Ελλάδα ξεκίνησε από μια πάρα πολύ χαμηλή αφετηρία στη χρήση γενοσύμων. Έχουμε ολοκληρώσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων στον τομέα τη υγεία και έχουμε εφαρμόσει μια σειρά μέτρων. Έχουμε ξεκινήσει να ανεβαίνουμε, ξεκινήσαμε από το 14% και τώρα πλησιάζουμε το 22%. Στόχος είναι στο τέλος του 2014 να φτάσουμε περίπου στο 60% χρήσης γενοσύμων φαρμάκων ε, στην ελληνική επικράτεια. Για να το πετύχουμε αυτό έχουμε ακολουθήσει μια πολιτική και μειώσεως της τιμής των γενοσύμων αλλά και παροχής κινήτρων φαρμακοποιούς για να ε, γράφουν γενώσιμα φάρμακα και βέβαια μια καμπάνια προς το κοινό, την οποία και σχεδιάζουμε, για να εμπεδώσουμε την αίσθηση ασφάλειας ως προς τα γενώσιμα φάρμακα. Γιατί εκεί υπήρχε μια ε, ας πούμε έτσι παρεξήγηση ε, στον ελληνικό πληθυσμό. Πάντως είναι βασικός άξονας πολιτικής μας η αύξηση της χρήσης των γενοσύμων φαρμάκων ως μέσο και ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης. Τώρα στο κομμάτι των ε, medical devices που θέσατε προηγουμένως, ε, το λέω και για την κυρία Ροντμπερντ, για την ελληνική προεδρία το φάκελος αυτός είναι ζήτημα μεγάλη προτεραιότητας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να το θέσουμε σε κίνηση και να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία όσο γίνεται ε, πιο γρήγορα, αντιλαμβανόμενοι τις μεγάλες διαφορές στην οπτική γωνία που τα διάφορα κράτη-μέλη ε, έχουν πάνω σε αυτό το ζήτημα. Όμως πιστεύουμε ότι το κοινό μας συμφέρον είναι να μην αφήσουμε μια τόσο μεγάλη εκκρεμότητα για το μέλλον. Και νομίζω ότι με αυτό το πνεύμα, σε πνεύμα ευρωπαϊκό, καλής θέλησης... θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά στο θέμα του DNA, ε, Όπω έχω πληροφορηθεί, το θέμα αυτό των εξάστων DNA έχει τεθεί στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου. Ε, δεν υπάρχει ακόμα τελική θέση και το θέμα αυτό εξετάζεται. Είναι πολύπλοκο ζήτημα και δεν είναι τόσο εύκολο να σα δώσω μια απάντηση. Ε, κυρία Ροντμπέρ, ξέρω ότι έχετε κάνει προσωπικά πολύ μεγάλη προσπάθεια για αυτό το θέμα. Και τη σέβομαι πάρα πολύ. Ε, γνωρίζω ότι υπάρχει από ορισμένε χώρε και υπήρξε μια κολυσιεργία ω προ προς το να προχωρήσει αυτό το ζήτημα μπροστά. Ε, πρέπει να σα πω ότι η ελληνική προεδρία ήδη το έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα. Έχουμε ήδη κάνει τα πρώτα θετικά βήματα. Τελειώσαμε την πρώτη ανάγνωση. 27-28 Ιανουαρίου έχουμε ομάδα εργασία για αυτό το θέμα και 11 και 12 Φεβρουαρίου. Πιστεύουμε ότι όταν θα ολοκληρωθεί η ομάδα εργασία, ομαδα εργασίας 11-12 Φεβρουαρίου θα είμαστε σε θέση να ας πούμε πολύ συγκεκριμένα σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και πόσο κοντύτερα έχουμε καταφέρει να φέρουμε τις θέσει των διαφόρων κρατών, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί. Ε, είμαστε απολύτως σύμφωνοι ότι όπως λειτουργεί σήμερα το σύστημα και με τα notified bodies και με το πώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα class, ή devices και όλα αυτά, ε, υπάρχει πρόβλημα και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα ε, και πρέπει να βρούμε εκείνο το σημείο ισορροπίας μεταξύ μιας ρυθμισμένης και ελεγχόμενης αγοράς που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την ασφάλεια των ασθενών που πρέπει να είναι ε, στην κορυφή όλης μας της συζήτησης από τη μια πλευρά χωρίς να χάσουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και τη δυνατότητα της ε, εξέλιξης από την άλλη. Πιστεύω ότι σε πνεύμα καλής θέλησης τώρα στην ερώτηση τι εξασφάλιση μπορούμε να έχουμε ε, <laughs> ότι όσο καλή διάθεση να έχω να σας πω εγώ ότι μπορώ να το εξασφαλίσω θα ήταν λίγο υπερβολικό εκ μέρους μου αλλά θέλω να ξέρετε ότι θα κάνουμε σε, σε πλήρες ευρωπαϊκό πνεύμα αυτό μπορούμε καλύτερα. Τώρα μια και αναφερθήκατε και εσείς μεταρρυθμίσεις θα μου επιτρέψετε και ένα προσωπικό σχόλιο ε, οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν τόσο γρήγορα. Και πιστεύω με επιτυχία, όπω θα πω και συνέχεια σε απαντήσει άλλων συναδέλφων, χωρί τη βοήθεια τη Task Force και προσωπικά του κ. Ράιχενμπαχ ο οποίος υπήρξε ε, πάνω από κάθε, κάθε βήμα αυτής της προσπάθειας με, με, όχι, με, ζέση πραγματική. Ε, αισθάνομαι ότι βρίσκεται στη χώρα μας και πονάει τη χώρα μας σαν να γεννηθεί σε αυτήν. Ε, προς την κυρία Τάιλε. Θα συμφωνήσω μαζί σας και πιστεύω ότι η πρόληψη είναι κλειδί στη μείωση των ε, βλαπτικών συνεπειών της κατάξυνο πνεύματος και θα πρέπει να εστιάσουμε στην προώθηση δράσεων αγωγή υγεία για το σύνολο του πληθυσμού με έμφαση στου νέου και στην πρόληψη των τροχαίων που αποδίδονται στο αλκοόλ. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει τον περασμένο Οκτώβριο την επεξεργασία στο πλαίσιο τη Επιτροπή Εθνικών Πολιτικών και Δράσεων, ΚΝΑΠΑ, ενό Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράση για τη μείωση των βλαβών από την κατανάλωση νοπνεύματο και η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται εντό του έτου. Αναμένουμε και εμεί το τελικό κείμενο. Ε, πρέπει να σα πω όμω ότι σε γενικέ γραμμέ η Ελλάδα δεν είναι χώρα που έχει τα περισσότερα προβλήματα στον τομέα. Έτσι, δεν είμαστε στην, στην πρώτη ταχύτητα. Ε, στον κύριο Χρυσόγελ. Θα τα πάω λίγο όπως, για, για, για να οργανώσω λίγο τη σκέψη μου. Στο θέμα της μετανάστευσης, στο οποίο θέσατε, ε, εμείς πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνονται απολύτως σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων και ούτε διανοούμαστε ως χώρα ότι θα αφήναμε του ανθρώπου ανυπεράσπιστου. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι για να τα καταφέρει η Ελλάδα ή και άλλε χώρε, οι οποίε δέχονται λόγω γεωγραφική θέσεω αυτά τα κύματα σε πρώτο χρόνο, δεν μπορούν να το κάνουν χωρί να έχουν τη βοήθεια και των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών. Εμεί λέμε ότι το ζήτημα τη μετανάστευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο στο πλαίσιο τη χώρα που δέχεται την πίεση, αλλά αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα γιατί όλοι οι Ευρωπαίοι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων και τη παροχή αυτού όλων των υπηρεσιών υγεία που κάθε άνθρωπο πρέπει να έχει. Όμω ε, η κάθε χώρα μόνη τη και φυσικά η Ελλάδα και οι παρούσε συνθήκε είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντέξει μόνη σε αυτό το φορτίο. Άρα χρειάζεται τη βοήθεια των υπολείπων Ευρωπαίων πολιτών, των υπολείπων Ευρωπαϊκών κρατών. Στο θέμα των ασθενειών ε, δεν είναι ακριβώ όπω το λέτε. Υπάρχουν ασθένειε που είχαν εξαφανιστεί στην Ελλάδα, θυματίω αναφέρθηκε και από επόμενο συνάδελφο, ε, ελενοσία, το τελευταίο διάστημα είχα μια πολύ μεγάλη ανησυχία και προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία για το θέμα τη πολιομελίτιδα, η οποία είχε κίνδυνο να έρθει από τη Συρία. Άρα δεν είναι αληθέ ότι δεν φέρνουν ασθένειε. Προφανώ φέρνουν, δεν του κατηγορώ γι' αυτό. Έρχονται από υποβαθμένε περιοχέ, καλύπτουν τεράστιε αποστάσει, προφανώ περνάνε από φοβερέ κακουχίε, άρα είναι πιο ευάλωτοι και πιο εκτεθειμένοι σε κινδύνου διαφόρων ασθενειών. Τώρα το ζήτημα δεν είναι να πούμε αν φέρνουν ή δεν φέρνουν. Προφανώ κάποιε φέρνουν, ίσω όχι στο βαθμό που κάποιοι θα θέλουν να το παρουσιάζουν. Το ζήτημα είναι πώ θα μπορέσουμε ω Ευρώπη, ω Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιμετωπίσουμε σωστά αυτό το φαινόμενο. Γιατί η διάδοση τέτοιου είδου ασθενειών, που παραμένω στην Ελλάδα ήταν εξαφανισμένε για 30 και 40 χρόνια, δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για την Ελλάδα, αλλά αποτελεί κίνδυνο και για την Ευρώπη. Γιατί διαδίδονται και μεταδίδονται. Άρα Εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο η ελληνική προεδρία θέλει να αναδείξει ούτω ή άλλω όλη τη διάσταση. Όπω να σα πω παραδείγματο χάρη ότι η παροχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσοκομιακή κάλυψη σε όλου αυτού του ανθρώπου την τελευταία δεκαετία έχει κοστίσει στην Ελλάδα εκατοντάδε εκατομμύρια. Και ξέρετε ότι η Ελλάδα θυμίζει μια θέση πάρα πολύ δύσκολη οικονομική και άρα κάθε ευρώ μετράει. Και ένα από τα σημεία στα οποία διάφορε, όπω είπα, τα ακροδεξιέ ομάδε ποντάρουν είναι στην οργή του πληθυσμού που δημιουργείται από την εντύπωση ότι ο πολύ φτωχό Έλληνα πληρώνει για αυτού. Ενώ δεν είναι άλλη θέση ότι είναι έτσι, αλλά έτσι προβάλλεται. Και αυτό δημιουργεί, ξέρετε, αντισυσπυρώσει στην κοινωνία που καλό να τι αντιμετωπίσουμε. Και όχι να τι αφήσουμε να υπάρχουν και να τι εκμεταλλεύονται κάποιοι για πολιτικού λόγου. Ε, στο θέμα του εμβολιασμού, πρέπει να σα πω ότι όλε οι μελέτε που έχουμε στα χέρια μα και του ΟΣΑ, η πρόσφατη έκθεση, αλλά και οι δικές μας ε, μελέτες δεν, ε, ε, καθόλου δεν επιβεβαιώνουν την εικόνα που κάποιοι θα προβάλλουν στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα ελλείψης εμβολιασμού ιδιαίτερα των παιδιών ή του πληθυσμού. Είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εν μέσω κρίση δεν έχουμε μειώσει καθόλου τα προγράμματα εμβολιασμού, ούτε κατά ένα. Και πέρσι το καλοκαίρι προέκυψε ένα πρόβλημα, μέσα από το Ινστιτούτο Παστέρ συγκεκριμένα. Ζητήσαμε το Γενικό Λογιστήριο και μα έδωσε έκτακτη χρηματοδότηση 3 εκατομμύρια ευρώ για να συνεχιστεί κανονικά το πρόγραμμα και να σταματήσει. Άρα δεν ισχύει. Η Ελλάδα δεν υπολείπεται των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών στο κομμάτι του εμβολιασμού. Ε, το κομμάτι της ε, υγείας και της κλιματικής αλλαγής είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ε, που ασφαλώς ε, θα άξω τον κόπο να επισημανθεί στην ελληνική προεδρία. Δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι, αλλά όντως το άξονα πολύ ενδιαφέρον όπως το είπατε. Παρόλο που η Ελλάδα στην παρούσα φάση της κλιματικής αλλαγής είναι ευνοημένη τρόπον την γιατί εμείς έχουμε ξέρετε μια παρατεταμένη περίοδο πολύ ποιον φαινομένων και το καλοκαίρι δεν είχαμε κάψουμε και το, το χειμώνα δεν έχουμε ε, πολύ μεγάλε έντονε πούμε έντονες ε, ε, καιρικές συνθήκες. Αυτό δεν λέει τίποτα. Προφανώ είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το παρακολουθούμε και μα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όπω το κομμάτι που είπατε για να οργανώσουμε κάτι σε σχέση με του πολίτε, με την κοινωνία των πολιτών, παρόλο που δεν το έχουμε στο πρόγραμμα, ε, θα σα απαντήσω και εγγράφω γιατί με ενδιαφέρει η ιδέα και πιστεύω να συνεργαστούμε το κάνουμε. Καθόλου δεν θα είχα αντίρρηση για κάτι τέτοιο. Ξέρετε, πολύ σωστά επισημαίνεται ότι υπάρχει όλη αυτή η μεγάλη κρίση η εικόνα και πάλι ότι 3 εκατομμύρια Έλληνε δεν έχουν πρόσβαση στα σήματα υγεία δεν είναι ακριβή. όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, πρόβλημα υπάρχει, αλλά δεν είναι ακριβή. Όλοι οι Έλληνε έχουν πρόσβαση στην νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν υπάρχει νοσοκομείο που θα διώξει άνθρωπο που θα πάει σε επίγοντα περιστατικά και θα πει: Έχω ανάγκη να το δεχτεί. Είτε είναι Έλληνε είτε είναι μετανάστε. Όλοι έχουν. Βεβαίω αυτό που δεν έχουν είναι στην καθημερινή περίθαλψη, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, στην παρακολούθηση των χρονίων νοσημάτων. Ε, ένα από τα κομβικά σημεία πάνω χάρη τη μεταρρυθμίσεω που κάνουμε τώρα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία σε συνεργασία με τον ΠΟΗ είναι η δημιουργία αυτού του δημόσιου συστήματο που θα έχει καθολική πρόσβαση. Δεν θα εξαρτά την είσοδο του ασθενού από το αν έχει ασφαλιστική κάλυψη ή όχι, αλλά θα μπορούν να μπαίνουν όλοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, στην κυρία Γιάννα Κουδάκη. Πρώτα απ' όλα να πω για του γιατρού που έρχονται στη Μεγάλη Βρετανία. Έχω και πολλού φίλου, η αλήθεια είναι, και πριν γίνει υπουργό και τώρα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει πάρα πολλού γιατρού. Ένα από τα προβλήματα του δικού μα συστήματο είναι ότι έχουμε 75.000 γιατρού. Για να καταλάβετε, στον πληθυσμό μα θα αναλογούσαν περίπου 25.000. Έχουμε πάρα πολλού γιατρού. Έχουμε πολλού ανθρώπου στην Ελλάδα που θέλουν να γίνουν γιατροί και έχουν γίνει καλοί γιατροί. Για να αξιοποιήσουμε όλου αυτού του γιατρού στην Ελλάδα θα έπρεπε όλο ο πληθυσμό να αρρωστήσει. Δεν είναι αυτό μια καλή ιδέα. Άρα κάποιοι γιατροί θα βρουν δουλειά και έξω. Το ότι βρίσκουν καλή δουλειά στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι κατά ανάγκη κακό για την Ελλάδα ούτε για αυτού. Πολλοί από αυτού μετά από κάποια χρόνια γυρίζουν στην Ελλάδα αφού έχουν κάνει μια μακρά περίοδο σε άλλη χώρα. Στη Μεγάλη Βρετανία αλήθεια είναι την προτιμούν σε ένα μεγάλο βαθμό και, και μετά στο δικό μα σύστημα υγεία και με πολλέ εμπειρίε. Δεν είναι, ξέρετε, εμένα ω Ευρωπαίο πια η ιδέα ότι μπορούμε να εργαζόμαστε σε διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε και να ανταλλάσσουμε μεταξύ μα αυτή την κινητικότητα τη εργασία δεν είναι κατά ανάγκη κακό πνεύμα. Είμαστε Ευρωπαίοι, είναι η νέα εποχή. Ε, πρέπει μόνο να σας πω ε, ότι στο κομμάτι των, ε, των μεταρρυθμίσεων και όλο αυτό το κομμάτι το οποίο τώρα κάνουμε εν μέσω κρίσης, το οποίο δεν ήταν εύκολο να γίνει, ήταν πάρα πολύ, πολύ σωστά είπατε γιατί ο λαός υποφέρει. Πράγματι υποφέρει σε ενεστώτα χρόνο, δεν υπέφερε σε παρελθοντικό χρόνο, υποφέρει και σήμερα. Όμως η Ελλάδα βίωσε μια τόσο μεγάλη κρίση που η ιδέα ότι θα μπορούσαμε σε ένα λεπτό να την ξεπεράσουμε χωρίς κανείς να να αισθανθεί τι συνέπειέ τη, νομίζω δεν είχε μεγάλη επαφή με την πραγματικότητα. Ελπίζουμε και η κυβέρνησή μα εργάζεται πάρα πολύ σκληρά για να κάνει αυτό το διάνυμα του χρόνου όσο γίνεται πιο σύντομο. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι ο κόμμα υποφέρει και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Αλλά μην νομίζετε ότι μπορεί να γίνουν και θαύματα. Αυτό εννοώ. Προσπαθούμε και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα, στον κύριο Τούσα. Κύριε συνάδελφε, ακούστε, Καταλαβαίνω την μεγάλη ιδεολογική διαφορά που έχουμε. Όμω θέλω να σα πω το εξή και μιλάω γενικά. Συνηθίζουμε πολλέ φορέ, όχι μόνο εσεί, γενικά, να επικεντρωνόμαστε στι αστοχίε που πιθανόν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει και λάθη και αστοχίε και προβλήματα. Αλλά ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο ωραιότερο τόπο του πλανήτη για να ζει κανεί. Παραμένει ο τόπο με την περισσότερη δημοκρατία παραμένει ο τόπο με, με τον περισσότερο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παραμένει ο τόπο που έχει δώσει τη μεγαλύτερη ευημερία στου πολίτε για πάρα πολλά χρόνια. Παραμένει ο τόπο που προωθεί την ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Το να πυροβολούμε διαρκώ την Ευρώπη και να την παρουσιάζουμε σε ένα είδο διαβόλου, με συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ άδικο για όσα έχουν επιτευχθεί όλε τι τελευταίε δεκαετίε με τη βοήθεια, τη συνδρομή και τον αγώνα πολλών ανθρώπων. Τώρα, στην Ελλάδα είχαμε πράγματι μείωση του προπολογισμού τη υγεία. Όμως να σας πω και συνάδελφε, ότι και το κόμμα σας, αλλά και διάφοροι άλλοι στην Ελλάδα, και πριν από μερικά χρόνια, όταν η Ελλάδα ξόδευε τα τριπλάσια χρήματα για την υγεία, ακριβώς τα τριπλάσια, αν ήμασταν εδώ, θα λέγατε περίπου τα ίδια. Μόνο που τότε τα ξοδεύαμε, γιατί τα σπαταλούσαμε και τα πετάγαμε δεξιά και αριστερά. Και διάφοροι θησάβριζαν εις βάρος του ελληνικού λαού. Όχι το κουκουέ. Δεν είπα ότι θησάβριζαν το κουκουέ. Είπα ότι διάφοροι άλλοι, αυτοί γύρω γύρω από τα κυκλώματα της υγείας. Σήμερα Έχουμε μειώσει πράγμα του προπολογισμού μα, όμω σε αυτό ακριβώ το σημείο έχουν συμβάλει μεταρρυθμίσει. Έχουμε μειώσει του προπολογισμού μα χωρί να μειώσουμε τι παροχέ υγεία στου πολίτε μα κατά καθόλου μάλιστα. Μπορώ δεν να σα πω ότι σήμερα τα νοσοκομεία μα έχουν λιγότερα ράτζα και δουλεύουν πολύ καλύτερα από ό,τι δουλεύουν από 5 χρόνια. Και το κάνουν αυτό με το 1 τρίτο των χρημάτων. Άρα μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Δεν είναι όλα μαύρα. Ε, και όπως είπα και πριν στον κύριο Χρυσόγελο, βασική μας, ε, βασική μας στόχευση στη μεταρρύθμιση πρωτοβάθμιου φροντίδας υγείας είναι να αποκτήσουν πρόβαση όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα ασφαλιστικής κάλυψης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. θα αρχίσουμε τώρα με το δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Θα δώσουμε το λόγο ε, σε μια νέα ομάδα ε, ανθρώπων, Πέτερλε, Στρέλα, ε, θα ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Α, και κάποιοι δεύτερη φορά, όπως η Ρεμπέκα Τέιλορ, βλέπω εδώ στον κατάλογο. Δεν νομίζω να ξέχασα κανένα, θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. Έχουμε ε, επίσης, ε, τι κάμερες βλέπετε, είναι από την ομάδα που έχει καλέσει η κυρία Χέμπνερ από το Πότστατ, ο κύριο Πέτερλε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ και να συγχαρώ και την ελληνική κυβέρνηση για την θετική αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Ως συμπρόεδρος ε, της ομάδας εργασίας για τα θέματα υγείας, και μέλος ε, της ειδικής ομάδας ε, των βουλευτών ε, που ασχολούνται με τις δράσεις καταπολέμησης του καρκίνου, χάρηκα όταν αναφερθήκατε στην αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας της Ελλάδας. Τρεις ερωτήσεις έχω να σας θέσω που εντοπίζεται μία ανάγκη να προσφέρουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μέσω δράσεων για την υγεία. Δεύτερον, ποια είναι τα βασικά στοιχεία της μεταρρυθμιστικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης. Ε, με λίγα λόγια, τι θα κάνετε για να ε, αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. λόγω τη κρίση χρειάζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και τρίτον, ποιε θα είναι οι δράσει κατά πολέμηση του καρκίνου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Επόμενη είναι η συνάδελφο Εστρέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, Ελληνιστή, λέει η κυρία Εστρέλα. Είμαι Πορτογαλίδα και παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή την κατάσταση στην Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τους Έλληνες που έχουν υποφέρει τόσο πολύ ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της πολιτικής λιτότητας, όπως και οι Πορτογάλοι. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για την Προεδρία σας. Υπουργέ, ήδη αναφερθήκατε στο ότι μία από τις προτεραιότητάς σας θα είναι να καταστήσετε βιωσιμότερο και αποτελεσματικότερο το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, βελτιώντας έτσι και την υγεία των πολιτών. Θα ήθελα να γνωρίζω τα συγκεκριμένα μέτρα που προτίθεται να παρουσιάσει και να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να υλοποιήσει αυτούς τους ε, προδιαγραφέντες στόχους. Ε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ζήτημα διότι ήμουν εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση σχετικά με την αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας και την μείωση των ανισοτήτων στον τομέα αυτό στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχέση με αυτά που είπατε, Υπουργέ, ότι στην Ελλάδα όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως έχουν ε, πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ξέρουμε ως αποτέλεσμα της κρίσης στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες αποκλείεται ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός πολιτών ε, που για οικονομικούς λόγους έχουν μειωμένο εισόδημα κατά 30% και ενίοτε και περισσότερο και ως εκ τούτου δεν έχουν ε, πρόσβαση σε απαιτούμενες ιατρικές υπηρεσίες ούτε και στην ε, ε, απαιτούμενη ε, φαρμακευτική περίθαλψη. Το 2011, βάσει στοιχείων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί του 3 έως 4% του ευρωπαϊκού πληθυσμού δεν είχε την ε, απαιτούμενη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας λόγω του κόστους, τη απόστασης και του μεγάλου παρατεταμένου χρόνου αναμονής. Αυτή η αρνητική τάση δεν πλήττει όλες ιδιαίτερα τι γυναίκε. Οι οικονομικές δυσκολίες ε, με ε, τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι πολίτες επηρεάζουν τις συνθήκες ζωής τους γενικότερα και ειδικότερα την υγεία τους. Θα κάνω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, Υπουργέ. Με ποιο τρόπο η ελληνική προεδρία θα συμβάλλει στην προσπάθεια αναστροφής αυτής της αρνητικής τάσης, αυτού του αρνητικού σεναρίου, αμβλύνοντας τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, στο εστερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ, ε, Ελληνιστή, κυρία Στρέλα. Σας ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Κουμουτσάκος έχει το λόγο. Thank you, treatment ευχαριστώ. Ελπίζω να μου δώσετε τον ίδιο χρόνο που δώσατε στους συναδέλφους της ενιαίας αριστεράς, λέει ο κ. Κουμουτσάκος. Επιτροπή Περιβάλλοντος, μια επιτροπή που έχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία ε, στα θέματα που χειρίζεται και ειδικότερα στα θέματα δημόσιας υγείας. Σας εύχομαι μια επιτυχημένη Προεδρία. Είναι μια απαιτητική Προεδρία. Αφενός γιατί συμπίπτει με τα τελευταία και γι' αυτό τα πιο επώδυνα βήματα εξόδου από την κρίση και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αφετέρου διότι λόγω των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών το νομοθετικό έργο που πρέπει να παράγει η Προεδρία συμπιέζεται στον περιορισμένο χρόνο των τριών-τεσσάρων μηνών. Επομένως, το, ο φόρτος εργασίας και η πίεση εργασίας θα είναι μεγάλη. Δεν θα αναφερθώ σε ζητήματα τα οποία έχουν θίξει οι άλλοι συνάδελφοι όσον αφορά την νομοθετική σας ε, ε, τον νομοθετικό σας προγραμματισμό. Όμως και εν ώψη και των ευρωπαϊκών εκλογών και του, του ιδιαίτερα ευαίσθητου πολιτικού χρόνου στον οποίο η Ελλάδα καλείται να ασκήσει τα καθήκοντα της Προεδρίας του Συμβουλίου θέλω να επαναλάβω και να επανέλθω σε μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας που αναφέρατε και αφορά τη σύνθεση δύο πολύ κρίσιμων ζωτική σημασία θεμάτων και ενδιαφέροντο για του Ευρωπαίου πολίτε. Μετανάστευση και δημόσια υγεία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συγχαρούμε την Ελληνική Προεδρία που ενέταξε αυτό το θέμα στι προτεραιότητέ τη. Γιατί αφορά και του Ευρωπαίου πολίτε και όπω είπαμε σε έναν πολύ ευαίσθητο πολιτικό χρόνο. Η μετανάστευση είναι αλήθεια ότι ασκεί μεγάλη πίεση στα ίδια επιβαρημένα συστήματα υγείας στην Ευρώπη και κυρίως στις χώρες του Νότου που δέχονται την, το οστικό κύμα αυτού του φαινομένου. Βέβαια η λύση δεν είναι ο αποκλεισμό των ταλαιπωρημένων και βασανισμένων συνανθρώπων μα από τα συστήματα υγεία. Αυτό είναι απολύτω ξένο και απορριπταίο από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ταυτόχρονα όμω δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μα σε μια πραγματικότητα. Η λύση δεν είναι η αδράνεια, δεν μπορεί να μείνουμε στην σημερινή κατάσταση χωρίς να δούμε ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Χρειάζεται λοιπόν ευρωπαϊκή λύση αλληλεγγύης. Τι εσείς, πέραν του ότι ανοίγετε αυτή τη συζήτηση ως Προεδρία και κάνετε πάρα πολύ καλά, μπορούμε να προσβλέπουμε ότι θα υπάρξει μια συμφωνία επί ενός πολιτικού κειμένου, πλαισίου, για το πώς ένα τόσο σύνθετο και δύσκολο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προφανώ ε, νομοθετικό έργο δεν μπορεί να παραχθεί διότι δεν έχει γίνει κάποια προεργασία. Αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμο, θα ήταν πολύ σημαντικό πέραν τη εκείνη τη συζήτηση, εάν εφόσον έχετε εντάξει αυτό το θέμα στι προτεραιότητέ σα, μπορέσουμε μέχρι το τέλο τη Προεδρία να έχουμε ένα κείμενο πλαίσιο αρχών ώστε να ακολουθήσουν με τη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη νέα Επιτροπή κάποιε νομοθετικέ πρωτοβουλίε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καλσλίτερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλώς ορίσατε Υπουργέ. Εάν έχουμε... Όχι, θα τα πω στα αγγλικά. Ε, αν έχετε πολλούς γιατρούς ε, θα έχετε και πολλές ΜΕΕΣ. Εμάς μας λείπουν οι ΜΕΕΣ. Άμα θέλετε να μας δώσετε μερικές, ευχαρίστως λοιπόν, ε, μιλήσαμε για την πολιτική για τα προϊόντα καπνού. Υιοθετήσαμε, ε, θα υιοθετήσουμε πολύ σύντομα τον νέο κανονισμό ε, και πιστεύω ότι εκεί δαπανώνται πολλά χρήματα για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, αλλά και για την σωστή υλοποίηση της νέας οδηγίας σε όλες τις χώρες. Για τους ενδοκρινικούς αναστολείς, ένα άλλο βασικό πρόβλημα ε, μιλήσαμε για τη δυσφενόλη και άλλες τέτοιες χημικές ουσίες. Ε, θα αναλάβετε πρωτοβουλίες ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, διότι θα βοηθούσε αυτό ώστε να ασκηθεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να επιταχυνθεί η δράση της. Νομίζω ότι ανάμεσα στην έκθεση και το αποτέλεσμα παρέρχεται ε, πολλής χρόνος και αυτό είναι μέλος, μέρος του προβλήματος. Ε, ως προς την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, υπάρχουν κάποια μέτρα, όπως η σήμανση, παραδείγματος χάρη των αλκοολούχων ποτών. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη παρανόηση στο κοινό ε, για την κατανάλωση του αλκοόλ, ε, τη σχέση με τον καρκίνο, ε, και σε σχέση με την σήμανση υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσει την πρότασή της του χρόνου. Τι πιστεύετε για τη σήμανση των αλκοολούχων γενικότερα. Αν και κάτι άλλο ε, σύντομο, ε, μιλήσατε και ο ίδιος για το κόστος των φαρμάκων Μιλήσαμε για την υποχρεωτική αδειοδότηση ε, και συζητήθηκε αυτό ως ενδεχόμενη λύση για κάποιες περιπτώσεις στην Ελλάδα αλλά και ως ένα καινοτόμο εργαλείο. Αντί να έχουμε δαπανηρά διπλώματα ευρεσιτέχνειας ε, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει πρόσβαση στα φάρμακα που ήδη υπάρχουν γιατί δεν έχει αρκετά χρήματα το κράτος για να τα αγοράσει, θα συζητηθεί ε, στην ελληνική προεδρία ένας καινοτόμος μηχανισμός για ένα εφάπαξε ποσό για καινοτόμα φάρμακα, δηλαδή η γνώση θα είναι δημόσια πλέον με το που κατασκευάζεται ένα νέο φάρμακο και καταβάλλεται το εφάπαξ αντίτιμό του, τότε όλες οι χώρες ε, στην Ευρώπη και στην Αφρική θα έχουν πρόσβαση και δεν θα πρέπει να περιμένουν 20 χρόνια για να ε, γίνει γενώσιμο το φάρμακο. Ε, προτίθεστε να συζητήσετε αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πολύ. ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτά που είπατε και για τα θέματα της αλληλεγγύης. Πράγματι είμαστε μια γενιά η οποία δεν γνώρισε τον πόλεμο και πολλοί ξεχνάνε το τι είχαν περάσει τότε οι άνθρωποι. Θα επανέλθω σε αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως κύριε Υπουργέ Αναφερθήκατε σε πολλά θέματα χωρίς υποχρεωτικά να προχωρήσετε σε βάθος ε, λόγω της ποσότητάς τους. Ένα από τα θέματα αυτά είναι η γύρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Γυράσκει ο ευρωπαϊκός πληθυσμός και θα πρέπει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο να προπαρασκευαστούμε σωστά έτσι ώστε αυτοί των οποίων το προσδόκιμο ε, ζωής μεγαλώνει να μπορούν να καλύπτουν τις ιατρικές τους ανάγκες. ιδιαίτερα στην πολύ μεγά, στις πολύ μεγάλες ηλικίε. Ε, γιατί θα φτάνουν όλο και περισσότερο σε τέτοιες ηλικίε οι πολίτες. Απαιτούνται λοιπόν προγράμματα κάλυψης των ιατρικών αναγκών ε, ισορροπημένα και διαρωτώ με αν προβλέπετε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες και το οποίο θα μπορούσε ε, να χρησιμεύσει σαν σημείο αναφοράς και εκκίνησης. Βέβαια φυσικά και λαμβάνοντας υπόψη ε, τα χαρακτηριστικά των επιμέρους χωρών. Κάποιες χώρες που έχουν πολλά μέσα μπορεί να εμβαθύνουν, κάποιες άλλες μπορούν να χρησιμοποιούν μια πιο light μορφή των προγραμμάτων αυτών. Το θέμα είναι λοιπόν να μην έχουμε για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου επιμέρους εθνικά προγράμματα, αλλά ένα βασικό ευρωπαϊκό. Σας ευχαριστώ. Άλλη μια ερώτηση από την κυρία Τέιλορ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ρωτώ εξ ονόματος του συναδέλφου Κρις Ντέιβις, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί εδώ σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να θίξω το θέμα της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη σύνδεση με τα προβλήματα τα αναπνευστικά αλλά και τα καρδιογειακά. Σήμερα το πρωί διάβασα μια έρευνα της BMJ σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες ε, που εξετάζει πάρα πολλά άτομα και επιβεβαιώνει αυτή τη σύνδεση μεταξύ της ρήπανσης της ατμοσφαιρικής και των καρδιακών παθήσεων. Αυτό που λέει το άρθρο η μελέτη είναι ότι η ποιότητα της ατμόσφαιρας και η νομοθεσία που διέπει έχει να κάνει, είναι εντό των. Ε, μάλλον δεν εγγυάται ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κατά πόσον θα κοιτάξει η Προεδρέα το θέμα τη ατμοσφαιρική ποιότητα, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια γενική αντίσταση στο θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Και τέλο, ο συνάδελφο Λάιε Πόκρου. κύριε Υπουργέ, και εγώ θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες οι οποίοι εξέφρασαν βασικά την αλληλεγγύη τους με τον ε, δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό ο οποίος εξακολουθεί να υποφέρει και θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι κυρίες και κύριοι <clears throat> γιατί έχει συμβεί αυτό. Μερικές φορές υπάρχει μια σύγχυση ε, ανάμεσα στη θεραπεία και στην διάγνωση. Δεν φταίει η θεραπεία, δεν φταίνε τα φάρμακα, αλλά δυστυχώς φταίει η ασθένεια που προκάλεσε την σημερινή κατάσταση. Αν δεν υπήρχε το πακέτο διάσωσης το οποίο δόθηκε από την Τρόικα και βασικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε θα είχε πτωχεύσει ξεκάθαρα η Ελλάδα και δεν θα είχε χάσει μόνο το 25% του ΑΕΠ αλλά το 50%. Λοιπόν, νομίζω ότι σε μια επιτροπή σαν τη δική μας που είναι γεμάτη ιατρικό προσωπικό πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο φάρμακο και την ασθένεια. Αλλά πέραν αυτού, αυτό το οποίο απαιτείται είναι η αλληλεγγύη. Λοιπόν, τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις. Η μία αφορά την συνεργασία με την Τουρκία. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία. Και δεν έχει καμία άλλη επιλογή νομίζω από το να συνεργαστεί με την Τουρκία σε τομείς όπως η δημόσια υγεία και σε θέματα που άπτονται φυσικά της μετανάστευσης κτλ και μιας και προεδρεύεται τώρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ίσως να μπορέσετε να μας πείτε πώς μπορεί η Ελλάδα να βοηθήσει την Τουρκία και αντίστροφα η Τουρκία την Ελλάδα στα προβλήματά τους. Δεύτερο θέμα είναι η επίπτωση της τραγωδίας στη Συρία. Είναι ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τους πρόσφυγες της Συρίας και την έβρεση πολιτικής λύσης. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει για να ελαφρύνει ε, την τραγωδία αυτή, ιδιαίτερα για τους πρόσφυγες υπάρχουν προβλήματα, ξέρετε, σε επίπεδο δημόσιας υγείας, υγιεινής ε, μεταδοτικές ασθένειες κτλ. Και τέλος, αναφερθήκατε στην ε, εκροή εγκεφάλων από την Ελλάδα προς τις άλλες χώρες. Δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα. Υπάρχει ισχύει και για χώρες όπως η Ρουμανία, όπως η Βουλγαρία και αυτές είναι δύο φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χάνουν τα καλύτερα στοιχεία τους. Υπάρχει μια τεράστια μετανάστευση εξειδικευμένου προσωπικού προς τη ΣΥΠΑ, προς τη Σουηδία και προς άλλες χώρες όπου τα επίπεδα αμοιβή είναι φυσικά ιδιαιτέρως υψηλά σε σχέση με τις χώρες προέλευσης. Μήπως μπορείτε να μας πείτε κάτι πώς θα βοηθήσετε τους Βούλγαρους γιατρούς, τους Ρουμάνους γιατρούς και τους Έλληνες γιατρούς να μείνουν στη χώρα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπρόκος και Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινάμε με τον ε, ε, κύριο Πέταλε. Ευχαριστώ πολύ για τις, ε, για τις ερωτήσεις. Ξέρετε, ε, στην Ελλάδα έχουμε πονήσει ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με την Task Force. Το ονομάζουμε Υγεία εν δράση. Το οποίο θα, θα έλεγα να το στείλουμε και στα mail όλων των μελών της Επιτροπής γιατί είναι ένα υπόδειγμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και πώς μπορούμε πράγματι σε συγκεκριμένους τομείς ε, το ένα κράτος να βοηθήσει το άλλο. Εκεί λοιπόν θα δείτε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που έχουν ξεκινήσει και άλλες που προβλέπεται να ξεκινήσουν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όπου ειδικοί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν έρθει στην Ελλάδα και μεταφέρουν τεχνογνωσία. Πρέπει να σπώ το κομμάτι της μετανάστευσης που ανέφερε προηγουμένως ο κ. Κουμουτσάκος. Εκεί χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και σε πρακτικό επίπεδο και όχι μόνο εμεί, αλλά πιστεύω όλε οι χώρε που είναι χώρε υποδοχή του μεγάλου μεταναστευτικού κύματο για να μπορέσει να γίνει η καλύτερη διαχείριση ενό θέματο που, όπω είπα και πριν, ε, αποτελεί ε, ευρωπαϊκό ζήτημα. Ε, στο Συμβούλιο, λοιπόν, θα προσπαθούμε να φέρουμε συμπεράσματα για να δείξουμε ακριβώ πώ μέσα στι συνθήκε κρίση η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μπόρεσε εμπράκτο να βοηθήσει μια χώρα σε κρίση όπω η Ελλάδα να κάνει το επόμενο βήμα μπρο. Και τέλος όσον αφορά τους ασθενείς και την πρόσβασή τους, που παραδείγματος πριν για, τον, για τους καρκινοπαθείς, εγώ δεν θα υποκριθώ ότι στην Ελλάδα είναι όλα ρόδινα, το αντίθετο, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, όμως ε, θα επαναλάβω ότι στις ε, εξαιρετικά ευάλωτες κατηγορίες ε, ανθρώπων, όπως με τους καρκινοπαθείς, δίνει το εθνικό σύστημα τα φάρμακά τους σε μεγάλο βαθμό εντελώς δωρεάν, ακριβώς για να μπορούν να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Και αυτό όχι εύκολα, γιατί έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα, όπω είμαι βέβαιος του γνωρίζετε. στην κυρία Αστρέλα. Μποντία. Ε, καταλαβαίνω ότι εμείς αυτή την, την κρίσιμη περίοδο της τριετίας οι δύο λαοί μας ε, βιώνουν κοινά προβλήματα. Ε, διότι η κρίση χτύπησε περισσότερο τις, τις δικές μας χώρες και έτσι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο συνέβη. Ε, πρέπει να σας πω ότι η ανισότητα στον τομέα της υγείας είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εγώ μάλιστα αύριο πρόκειται να μιλήσω ε, ε, εδώ σε μια ειδική ημερίδα για το θέμα των ανισοτήτων. Θα πρέπει να σας πω ότι υπό την προεδρία του Σερ Μάικλ Μάρμοτ φτιάχνεται το, το ειδικό δίκτυο ε, με έμφαση για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και πώς θα καλυφθούν αυτές οι κοινωνικές ανισότητες στον τομέα της υγείας. Έχουμε προσπαθήσει αυτή την περίοδο τη κρίση να βάλουμε στην πατρίδα μα πρακτικά θέματα τα οποία θα μειώσουν αυτές τις ανισότητες. Παραδείγματο χάρη, φτιάξαμε το λεγόμενο voucher για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, όπου μεταφέρουμε πόρου από ευρωπαϊκά προγράμματα και παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίε πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία σε ανθρώπου οι οποίοι έχουν μηδενική ασφαλιστική κάλυψη ή πολύ χαμηλό εισόδημα. Ακριβώ για να μην παραμένουν αποκλεισμένοι από υπηρεσίε που μπορούν να απολαμβάνουν άλλοι οι οποίοι έχουν καλύτερα εισοδήματα. Σε κάθε περίπτωση, κατά διάρκεια τη Προεδρία μα, προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο και είναι ένα από τα τμήματα για τα οποία συνεργαζόμαστε και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, ο οποίο μα μεταφέρει και τι δικέ του εμπειρίε, πώ μπορούμε να φτιάξουμε ένα ελάχιστο, όπω το λέμε, health safety net, ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών υγεία για του πιο αδύναμου, όπου τα κράτη-μέλη και η Ελλάδα πρώτα απ' όλα θα παρέχει σε όλου του ανθρώπου για να μειώσει αυτέ τι ανισότητε. Δεν υποκρίνομαι, παραλαμβάνω ότι όλα πηγαίνουν καλά. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, γιατί ναι, μεν ε, στα επίγοντα περιστατικά όλοι έχουν πρόσβαση και δεν αρνούμε σε κανέναν τη θεραπεία, αλλά στην καθημερινή φροντίδα οι άνθρωποι που έχουν χάσει την ασφαλιστική του κάλυψη, οι άνεργοι, είναι σχεδόν αποκλεισμένοι. Και όλη η μεταρρύθμιση την οποία κάνουμε τώρα και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία γίνεται για να μπορούμε να δώσουμε πρόσβαση σε αυτού του ανθρώπου. τώρα, ε, στον κύριο Σκλάιτερ. Σκλίτερ, okay για τη σήμανση των αλκοολούχων ποτών, που εγώ προσωπικά δεν είμαι αντίθετος, ε, είναι ζήτημα και άλλων Υπουργείων και των, ε, που έχουν να κάνουν με τα τρόφιμα. Ε, εμείς είμαστε περισσότερο στην πρόληψη εστιάζει του Υπουργείου Υγείας παρά στο κομμάτι της σήμανσης. Ε, φαντάζομαι ο συνάδελφό μου που θα ακολουθήσει, ο κ. Σαφθαρής που έχει την αρμοδιότητα, αν του κάνει σχετική ερώτηση να μπορεί και να απαντήσει πιο συγκεκριμένα. Πάντως εγώ προσωπικά ε, είμαι υπέρ μια τέτοια ε, μεταρρύθμιση. Ε, τώρα όλο το κομμάτι α, της μεταρρύθμισης στο κομμάτι της, ε, των νέων φαρμάκων και της πατέντας και το πώς θα μπορούσε να γίνει κτήμα στην παγκόσμια γνώση με πολύ ενδιαφέρον το άκουσα, φιλομολογήσω. Δεν έχουμε κάνει κάτι γι' αυτό. Ε, Εμεί κινούμαστε περισσότερο μέσα από τη συμφωνία, της Κλινικές δοκιμέ και αν θέλετε πιο ορθόδοξους, δρόμου, δρόμους, να το πούμε έτσι. Ε, καταλαβαίνουμε σε αυτό το οποίο είπατε. Ίσως θα ήταν μια λύση που θα μείωνε τις ανισότητες σε επίπεδο πλανήτη πια, αλλά καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι πιο σύνθετο ζήτημα. Για την άλλη, έχει κάποιε μηχανίε που επενδύουν πάρα πολλά χρήματα για να φτιάξουν ένα καινούριο φάρμακο και δεν ξέρω πώ μπορεί να, πώς να κάνει μια τόσο μεγάλη μεταβολή. Ε, Πάντω είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Θα άξιζε τον κόμμα να συζητηθεί εν για το πώ θα μπορούσε να γίνει. Δεν είναι θέμα τη ε, ελληνική προεδρία. Ε, στον ε, κύριο Κουμουτσάκο. Ε, κύριε Σνάλφε νομίζω θέσατε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Η Ελλάδα και πιστεύω και η Ιταλική Προεδρία που θα ακολουθήσει γιατί συνεργαζόμαστε το ίδιο πρόβλημα ως, ως χώρες υποδοχής αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πραγματικά ζήτημα. Ένα ζήτημα που δεν θα μπορούσε να εντοπιστεί σε επίπεδο χωρών παρά μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και όπω πολύ σωστά είπατε, ο Ευρωπαϊκό Πολιτισμό δεν θα άφηνε ποτέ σε κανένα μα να αρνηθεί υπηρεσία υγεία υγείας σε όποιον άνθρωπο τι έχει ανάγκη. Άλλωστε γι' αυτό είπα πριν ότι η Ευρώπη παραμένει ο καλύτερο τόπο για να ζει κανεί, γιατί έχουμε ακριβώ αυτέ τι αξίε, όπου άλλα μέρη του πλανήτη μπορεί να μην είναι αυτονόητες, σε εμά όμως είναι. Άρα το ζητούμενο είναι πώ θα μπορέσουμε αυτό το πρόβλημα που την λάβει διαστάσεις ορισμένε χώρε, στην Ελλάδα έχει λάβει σίγουρα θα μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σίγουρα στα συμπεράματα του δικού μας Συμβουλίου θα μπει αυτό το θέμα, γιατί νομίζουμε ότι αν μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε και να οργανώσουμε την κοινωτική ελεγγύη σε τον τομέα, θα έχουμε πραγματικά πολύ καλύτερα αποτελέματα και για τις χώρες υποδοχής και για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έρχονται και οι οποίοι πρέπει να έχουν μια ανθρώπινη αντιμετώπιση. Και αυτό είναι ο στόχος της Προεδρίας μας. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε δίνουμε στην κυρία Χίμπνερ. Ε, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια στην αρχή. Πρέπει ε, να ξέρετε ότι η κυβέρνησή μας κάνει, σας, σας το ανθρωπίνως δυνατό υπό δύσκολες συνθήκες, όχι εύκολες. Εγώ δεν εύχομαι σε καμία χώρα και σε καμία κυβέρνηση να μην περάσει τη δοκιμασία που έχει περάσει η Ελλάδα τελευταία χρόνια δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη γύρανση του πληθυσμού. Η Ελλάδα είναι μία από τι χώρε που αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Και πρέπει να σα πω ότι είναι λίγο σαν τον γόρδιο δεσμό που έκοψε ο μέγα Αλέξανδρος σε μία πόλη μικρά Ασία πριν από 2.500 χρόνια περίπου. Γιατί συμβαίνει το εξή. Ο πληθυσμό γυράσκει, άρα οι ανάγκε για υπηρεσίε υγεία αυξάνονται, άρα και το κόστο αυξάνεται, αλλά από την άλλη οι εθνικοί προπολογισμοί για τα συστήματα υγεία μειώνονται. Και δεν μειώνονται μόνο στι χώρε με μνημόνιο, όπω η Ελλάδα, μειώνονται σε όλε τι χώρε. Άρα λοιπόν πρέπει να συνδυάσουμε δύο αποκλίνουσε μεταξύ του καταστάσει. Πιστεύω όμω ότι δεν έχει άλλη λύση η Ευρώπη παρά να το κάνει και σίγουρα θα συμφωνήσουμε μαζί και θα το θέσουμε και στην Προεδρία μα ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα παρά σε, ε, σε επίπεδο τη κάθε χώρα μέλου ξεχωριστά. Γιατί όντω η υγεία του πληθυσμού είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα στην κυρία Τέιλορ για τον κύριο Ντέιβις είναι η ερώτηση. Ε, ασφαλώς και το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Εμείς το ξέρουμε στην Ελλάδα για πολλούς λόγους. έχουμε αντιμετωπίσει ως ατμοσφαιρική ρήπανση στην πρωτεύουσα τη του 80 λόγω των αυτοκινήτων. Το αντιμετωπίζουμε τώρα λόγω του προβλήματος στην θέρμανση των οικειών σε ορισμένε μέρες. Ε, έχουμε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Ε, να πω ότι πρωτοβουλίες για αυτό το θέμα ανήκουν περισσότερο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος παρά στο Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας ε, στην Ελλάδα έχει επισημάνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι από την επιβάρυνση της ε, ατμοσφαιρικής ρήπανσης για τη δημόσια υγεία και ε, ζητάμε σχεδιασμό συνολικής πολιτικής για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Σίγουρα θα πρέπει να απασχολήσει την Ευρώπη. Ε, δεν είναι πρόβλημα μόνο ελληνικό, είναι πρόβλημα σε διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε. Τέλο τον κύριο Μπόκρο. Θα συμφωνήσω απολύτω μαζί σα ότι χωρί το πακέτο βοήθεια η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν πολύ χειρότερη. Άλλωστε γι' αυτό ψήφισα όλα τα προγράμματα τα οποία τέθησαν προ ψηφοφορία έχοντα απόλυτη συνείδηση ότι αν δεν είχαμε την, ε, το πακέτο αυτών χρημάτων σήμερα η Ελλάδα θα είχε ήδη καταστραφεί. Αυτό πολλοί συνάδελφοί μου δεν μπορούν να το καταλάβουν και πολλοί Έλληνε το καταλάβουν ακόμα, αλλά δυστυχώ είναι μια πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει χάσει τώρα το 25%. Εάν είχε χρεοκοπήσει δεν θα είχαν το 50%, θα είχαν το 70% του εισοδήματό τη και σήμερα θα, ήταν, ε, θα θύμιζε χώρα όπω Σαχάρη Αφρική. Αυτό δεν έχει συμβεί χάρη στη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία και αναγνωρίζουμε. Από την άλλη όμω, γιατί όλα τα νομίματα έχουν δύο όψει, ε, θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι αυτό δεν έγινε χωρί τεράστιε θυσίε από του Έλληνε και χωρί πολύ μεγάλη πίεση. Μόνο να σα πω ότι η ανεργία στην Ελλάδα σήμερα είναι στο 27%. Είμαστε η πρώτη χώρα τη ανεργία στην Ευρώπη. Η δε ανεργία στου νέου αγγίζει το 60%. Άρα καταλαβαίνετε δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε την οικονομία μα, γιατί αλλιώ θα έχουμε χάσει μια ολόκληρη γενιά. Και αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνει και είναι και ένα, αν θέλετε, ευρωπαϊκό στοίχημα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα, τα ειδικότερα θέματα που θέσατε με την Τουρκία και τη μετανάστευση, παραδείγματο χάρη. Καταρχά η Ελλάδα συνεργάζεται με την Τουρκία. Ασφαλώ είμαστε γείτονε με την Τουρκία και κανένα μα δεν πιστεύει ότι θα έχουμε μέλλον χωρί συνεργασία και με την Τουρκία, που είναι ο βασικό μα γείτονα. Ασχέτω των όποιων άλλων προβλημάτων μπορεί να έχουμε, σα θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει ανοιχτά ζητήματα. Υπάρχει κατοχή στην Κύπρο, την οποία δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και την οποία θα πρέπει να βοηθήσουμε επίση. Πέραν όμω αυτών των ζητημάτων, τα οποία δεν ξεχνάμε, συνεργασία με την Τουρκία υπάρχει σε διάφορα επίπεδα και στον τομέα της υγείας ιδιαίτερα. Ε, το νέο πρόγραμμα έρευνας Horizon 2014-2020 ε, δίνει πολλές δυνατότητες με, στην Ελλάδα και στην Τουρκία καθώς και με τις άλλες χώρες των Βαλκανίων. Για το κομμάτι μετανάστευση να σας πω ότι μέχρι στιγμής η Τουρκία δεν είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμη για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς μεταξύ μα. Η Τουρκία έχει υπογράψει διάφορες συμφωνίες και με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επανεισδοχή των μεταναστών που έρχονται το δικό του έδαφο, τι οποίε πραγματικότητα υπογράφει αλλά αρνείται να εφαρμόσει. Και αυτό είναι κάτι που να, απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι συμφωνίε που υπογράφουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι οποίε δεν τηρεί. Και νομίζω εμεί οι Ευρωπαίοι μπορούμε να, να καταλήξουμε και να συμφωνήσουμε ότι εδώ στην Ευρώπη ισχύει το αρχαίο λατινικό ρητό Pacta sunt servanda. Άμα υπογράφει μια συμφωνία πρέπει να τηρείται. Η Τουρκία δεν τη στηρεί στο συγκεκριμένο θέμα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα στο κομμάτι της, ε, των γιατρών και γενικά του εξειδικευμένου προσωπικού που φεύγει από τις χώρες. Υπάρχει ένα joint action πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όπου προσπαθεί να θέσει κάποιο κίνητρα για την αναστροφή αυτής της τάσης. Εγώ δεν θέλω να υποκρίνομαι, μου αρέσει να μιλάω πιο πολύ στον πραγματικό κόσμο, όσο η ενεργεία είναι μεγάλη στις χώρες που αναφέρατε και η διαφορά των μισθών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή ήταν ένα γιατρό στην Ελλάδα μπορεί να μείνει άνεργο 2, 3 και 4 χρόνια. Και αν καταφέρει να βρει δουλειά, θα έχει ένα μέσο εισόδημα τη τάξη των 2.000 ευρώ το μήνα. Ενώ μπορεί να πάει στην Αγγλία και να βρει δουλειά με 6.500 λίρε το μήνα, πρέπει να σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον πείσει να μείνει. Δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. διότι έτσι δουλεύει η ελεύθερη αγορά. Και αυτή είναι η βασική τη ιδέα. Σε κάθε περίπτωση πάντω, την ελληνική κυβέρνηση να απασχολεί το ζήτημα κυρίως της απώλειας εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Γιατί, γιατί πραγματικότητα οι χώρες μας, όπως αναφέρατε η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, επενδύουμε χρήματα για να εκπαιδεύσουμε κάποιον να αποκτήσει κάποιες μεγάλες δεξιότητες, αλλά τελικά η ίδια η χώρα δεν κερδίζει αυτή την επένδυση, γιατί η επένδυσή της πιάνει τόπο σε μια άλλη χώρα. Και άρα αυτό είναι ένα υπαρκτό ζήτημα που απασχολεί και την ελληνική προεδρία και σίγουρα πρέπει να απασχολεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ Γεωργιάδη για την παρουσίαση αυτή. Θα πρέπει να πω ότι χαίρομαι και ανυπομονώ για τη συνεργασία μας τους επόμενους μήνες και χαίρομαι ιδιαίτερως που η Ιρλανδία Ε, πρόκειται για μια χώρα που έχει την προεδρία που ε, έχει παράδοση στη δημοκρατία. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, δυσκολίες, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα υπερβληθούν αυτές οι δυσκολίες. Και ξέρω ότι πολλοί πολίτες έχουν υποφέρει τα πάντα, να έχουν κάνει πάρα πολλές θυσίες και πιστεύω σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να μην χαθεί μια ολόκληρη γενιά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τεράστια η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Δεν θα πρέπει να το δάκτυλο δικτούμε ο στον άλλον, όχι. Να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί το πρόβλημα και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας είναι μεγάλη η ευθύνη μας, γιατί μόνο μία υγεία, μόνο ένα σώμα έχει ο καθένας μας. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν μπορούμε να βελτιώσουμε λοιπόν όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στον κλάδο αυτό, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και εκτός αυτού, αυτό που μου άρεσε πολύ είναι ότι πολύ συχνά ε, παραπονιούμαστε από πολύ ψηλά είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, ομολογουμένως, αλλά είμαι απόλυτα βεβαίως ότι από κοινού με αλληλεγγύη θα βγούμε από την κρίση και θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις σας. Εύχομαι ότι καλύτερο, ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσίασή σας. Συγχαρητήρια. Και νομίζω ότι μίλησαν πιο πολλοί συνάδελφοι και όλοι σας καλωσορίζουμε εδώ στην Επιτροπή και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση των μεμονωμένων φακέλων θα καταφέρουμε ε, εδώ στο Κοινοβούλιο να τα ξαναπούμε. Δεν είμαστε κυβέρνηση, είμαστε βουλευτές. Γι' αυτό λοιπόν και είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.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 Να παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους να ξανακαθίσουν στις θέσεις τους, παρακαλώ. Και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Και τον συνάδελφο Σλούτερ. Τη συνάδελφο Ροντ Μπέρεντ. Mhm. Yellow card. Äh, dass wir jetzt beginnen. Να ξεκινήσουμε, αν θέλετε. Έχουμε μια ένσταση βάσει του άρθρου 88 σε ό,τι αφορά την χώρα καταγωγής και την προ προέλευσης ε, κρέατος. Έχουμε κάποιους συναδέλφου εδώ που συνυπέγραψαν την ένσταση αυτή. Να δώσω στον κύριο Σλούτερ, στην κυρία Λιετάρτ, στην Σοφία Κονή, το λόγο. Πρώτος, πρώτη η Γκλένις Βιλμούτ. I didn't, I didn't Ναι, συγγνώμη, δεν άκουσα τι είπατε, Πρόεδρε. Είναι απίστευτο ότι κάνουμε καν αυτή τη συζήτηση. Το Κοινοβούλιο πάντα ήταν υπέρ της επισήμανσης της χώρας καταγωγής και του τόπου προέλευσης και του τόπου σφαγής και αυτό το ζητούν και οι ομάδες καταναλωτών ακόμα και οι ΙΠΑ πλέον ε, αναφέρουν τον ε, τόπο προέλευσης και σφαγής και θα σκεφτόταν κανείς ότι τουλάχιστον το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου θα έσπερχνε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει μεγαλύτερη διαφάνεια. Και πολλά κράτη-μέλη το ζήτησαν όταν ξέσπασε το σκάνδαλο. Φυσικά θέλουμε να υπάρχει τέτοια αναφορά του χώρου προέλευσης, χώρου προέλευσης και για το μεταποιημένο κρέας. Θα επανέλθουμε σε αυτό, αλλά θα πρέπει καταρχάς να τελειώσουμε και να ολοκληρώσουμε τους βασικούς κανόνες η επισήμανση του τόπου σφαγής και της χώρας προέλευσης επιτρέπει στον καταναλωτή να δει από πού έρχεται το κρέας, πόσο έχει ταξιδεύσει και να κάνει την αναλογή επιλογή. Οι καταναλωτές έχουν ήδη ε, συνηθίσει για το βόλιο κρέας αυτό το σύστημα επισήμανσης γιατί δεν υπάρχει διπλό σύστημα για άλλα είδη κρέατος. Και αυτό είναι παραπλανητικό και είναι κατά της νομοθεσίας να λέμε ότι ένας χείρος έχει έκτραφει ε, σε μια χώρα όταν ε, έχει ζήσει μόνο ένα ή τέσσερις μήνες ε, σε αυτή τη χώρα. Είναι ε, παραπλανητικό αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να καταργηθούν αυτές οι εξαιρέσεις σε ό,τι αφορά και τα συστατικά σε λουκάνικα, σε μεταποιημένο κρέα. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει την θέση της. Ξέρω ότι μεταμετωπίζει μεγάλη πίεση από κάποια κράτη-μέλη, από τον κλάδο τον μεταπητικό, αλλά δεν είναι αποδεκτή αυτή η λύση ούτε για το Κοινοβούλιο, ούτε για τους καταναλωτές. 83% των καταναλωτών δηλώνουν ότι θέλουν αυτές τις πληροφορίες και ότι είναι απαραίτητο αυτό το βήμα για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βέλμουτ. Καρμ Σλούτερ, επόμενος. Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Βίλμοτ, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά αρνήθηκε να μειώσει το χρόνο μεταφοράς για τα ζώα. Και αν έχουμε την αρχική σήμανση και για τους τρεις τόπους, ε, ο μας επιτρέπει ως καταναλωτές να γνωρίζουμε ε, το αν έχει υποστεί τρεις μεταφορές ε, διαφορετικές από την αρχή της ζωής του. Ε, εάν δεν υπάρχει αυτή η σήμανση θα αγνοούμε την ύπαρξη δύο μεταφορών. Σε σχέση τώρα με τη σήμανση βοήου έχουμε και τους τρεις τόπους και αυτό θέλαμε να αντιγράψουμε και να μεταφέρουμε. Λοιπόν στην αξιολόγηση αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν είναι ρεαλιστικός ο, ο υπολογισμό κόστους. Αντί να έχουμε σε ένα από τα παραδείγματα 10% αύξηση κόστους, παραδείγματος χάρη, και να απορρίψουμε αυτή τη λύση, εξακολουθούν να την προκρίνουν κάποια κράτη-μέλη. Ξέρουμε όλοι ότι η τιμή του βοηού δεν έχει αυξηθεί κατά 10% διότι εδώ ζούμε και το γνωρίζουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο μεγαλύτερο το κόστος για άλλα είδη κρέας. Εντάξει, για τα πουλερικά μπορώ να το καταλάβω, αλλά σίγουρα δεν φτάνουμε σε ποσοστό 10%. Είναι ψευδές το ποσοστό ε, και χρησιμοποιείται ως πρόφαση για να ε, κερδίσει την υποστήριξη των κρατών μελών. Στη συνέχεια μιλάμε για τα μεταποιημένα προϊόντα κρέατος. Ε, είναι ακόμη πιο περίπλοκη η κατάσταση. Αν έχετε 10% κρέας μέσα σε μία πίτσα, παραδείγματος χάρη, και λέτε ότι η πίτσα θα κοστίζει 10% ε, παραπάνω, τότε σημαίνει ότι διπλασιάζεται η τιμή του κρέατος. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό. Ε, μιλάμε για κομμάτια κρέατος ε, και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την άποψη των καταναλωτών που είναι υπέρ της τριπλής σήμανσης ε, παρότι αυξάνει το κόστος. Γιατί δεν κάνετε αυτό που θέλουν οι καταναλωτές, ε, αυτό που θέλει το κοινοβούλιο και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Αν έχετε παράπονα από τη βιομηχανία και αυτό σας ενοχλεί να μας το πείτε. Σας ευχαριστώ πήρα να τα Ναι, συγγνώμη ήμουν αφηρημένη. Εγώ είμαι κατά της, ε, του ψηφίσματος αυτού και να σας πω γιατί. αναφέρεται σε κάτι το οποίο συνέβη σε ό,τι αφορά τη σήμανση και σε ό,τι αφορά τον κανονισμό της σήμανσης. Είχαμε συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθέσει μία μελέτη αντικτύπου για τη σήμανση χώρας προέλευσης για τον οπόκρεας για να ξέρουμε κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό, τι κόστος συνεπάγεται και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να προβεί σε μια ρύθμιση σε ό,τι αφορά τον Αυτό λοιπόν και το έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποπίεση χρονική, το ομολογώ, γιατί η μελέτη που ξέρετε παίρνει και χρόνο δεν ήμουν και τόσο ενθουσιασμένη από το γεγονός ότι δεν υπήρξε μια πρώτερη ενημέρωση. Ευνηδιαστήκαμε ως Επιτροπή σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για την επισήμανση νοπού κρέατος. Αλλά στην τελική ανάλυση ήταν μια αρκετά σωστή ρύθμιση η οποία στέκει ελέγχθηκε κατά πόσον υπάρχει πραγματικά μεγάλο συμφέρον για τον καταναλωτή να υπάρχει αυτή η σήμανση του νοπού κρέατος, γιατί αυτό ήταν πάντα η, αντίπο, η εντύπωση που επικρατούσε. Και ρωτήσαμε λοιπόν τον καταναλωτή, τι θέλεις να επισημανθεί. Ο καταναλωτή λέει ναι, ναι, ναι, όλα, ό,τι έχετε δώστε μας. Αν ρωτήσουμε όμως τον καταναλωτή κατά πόσον είναι σε... προτίθεται να πληρώσει και για αυτή την επιπρόσθετη επισήμανση, ε, τότε λίγο αποτραβιέται, λίγο ε, διστάζει ο καταναλωτής και μας λέει «Α, όχι και έτσι, αν είναι να πληρώσω και άλλα χρήματα, δεν με ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση η επιπρόσθετη επισήμανση». Αυτό συμβαίνει λοιπόν. Αυτό συμφέρει 10% τους καταναλωτές μόνο. 40% των καταναλωτών αναφέρει ότι ούτε καν προσέχει την επισήμανση προέλευσης ε, στα καταστήματα. Αυτό το λέει και η έρευνα των οργανώσεων του καταναλωτή. Και καταλαβαίνετε, αν αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, φανταστείτε ποια είναι και τα πραγματικά στοιχεία. Γιατί οι καταναλωτέ ε, προφανώ αναφέρουν και ωραιοποιούν λίγο τα πράγματα. Όλοι οι καταναλωτέ είμαστε και τα γνωρίζαμε. Είμαστε δύσκολοι, ξέρετε, του καταναλωτέ. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι τόσο συντριπτικό είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον των ε, καταναλωτών για την σήμανση χώρος προέλευσης. Αυτό το διαπίστωσε και η μελέτη αντικτύπου. Τέταρτο λοιπόν ε, είναι το ενδιαφέρον. Καταρχάς πρώτον ενδιαφέρον είναι η ασφάλεια, δεύτερον ε, η γεύση, τρίτο ε, η τιμή και τέταρτο είναι μόνο η προέλευση του κρέατος. Και φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα στον καταναλωτή κατά πόσο προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι το κρέας. Και αυτό λοιπόν μέτρησε για την επισήμανση και για τη σχετική απόφαση. Οι δυνατότητες τώρα για την επισήμανση ε, έχουν διαφορετικό κόστος, προφανώς. Για την εκτροφή και το, τη σφαγή, εάν υπάρχει λοιπόν διπλή τέτοια αναφορά, και αυτό φαίνεται ότι απασχολεί τους καταναλωτές, είναι και η πιο ευνοϊκή ρύθμιση αν υπάρχει και η γέννηση και η εκτροφή και η σφαγή, αυτή η τριπλή αναφορά, αυτό συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερο κόστος και διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις μεταξύ 20-130.000 ευρώ παραπάνω ανά έτος. Είναι τεράστιο το κόστος θεωρώ. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις, μιλάμε και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται για τις αρχές. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την παρακολούθηση του συστήματος και αυτό έχει τεθεί και στο, στη συζήτηση για την ασφάλεια των τροφίμων. Κατά πόσον τα κράτη-μέλη προτίθενται να επενδύσουν τόσα χρήματα για τους έλεγχους αυτούς. Για τον καταναλωτή ασφαλώς υπάρχει και ο Πρόεδρος ε, καλεί την κυρία Ζόμερ να ολοκληρώνει. Ναι, ναι, ολοκληρώνει. Η δεύτερη ε, εναλλακτική είναι φυσικά συμφέρει πιο πολύ από οικονομικής άποψης γιατί τελικά το κόστος το πληρώνει ε, ο καταναλωτής. Σας παρακαλώ λοιπόν να καταψηφίσετε την πρόταση αυτή. Κύριε Ντοκμέρεν, σε πέντε λεπτά θα έρθει και ο Υπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, μου κάνει εντύπωση που όταν ακούω την ε, κυρία Σόμερ, γιατί η κυρία Άιγνερε που ε, δεν είναι πλέον υπουργό, είχε πει ότι φυσικά πρέπει να ξέρουμε τον τόπο προέλευσης ε, πρέπει να ξέρουμε αν γεννήθηκε εκεί το ζώο ή εξετράφει εκεί, αλλά και πάλι πέρα από όλα αυτά Πιστεύει κανείς ότι ο καταναλωτής ενημερωμένος ή όχι μάθει ότι ε, έγινε η εκτροφή για τέσσερις μήνες σε ένα συγκεκριμένο μέρος, ε, δεν μπορεί να ε, χαρακτηριστεί αυτό ως τόπος εκτροφής. Όλοι θέλουν να ξέρουν από πού είναι το ζώο, πού γεννήθηκε. Και όλα αυτά ξεκίνησαν με την όσο των ε, τρελών αγελάδων. Όλοι ήθελαν να ξέρουν ε, ε, πού γεννήθηκε το ζώο, από πού ήταν το συγκεκριμένο βόδι. Και εν πάση περιπτώσει λέτε ότι δεν θέλει να πληρώσει ο καταναλωτής γιατί θα είναι πιο ακριβό με τη σήμαση. Δεν το έχει αποδείξει ποτέ κανείς αυτό και πραγματικά ε, είναι ε, ντροπή αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραπέμπω στο άρθρο 26. Ε, λέει το άρθρο 26 ένδειξη τόπου γέννησης ή τόπου προέλευσης πρέπει να είναι υποχρεωτική. Με κάποιες εξαιρέσεις. Γιατί χρησιμοποιείτε τις εξαιρέσεις αναρωτιέμαι και γιατί βγάζετε και τα υπόλοιπα, τα κατάλοιπα κρέατος ε, και το, το κοιμά από αυτό, γιατί ε, εφαρμόζετε τέτοιες εξαιρέσεις. Μπορώ να σας πω, ξεκαθαρίσω ότι θα βγάλω ανακοινωθέν τύπου στη Γερμανία και θα εξηγήσω ποιοι είναι αυτοί που θα της να είναι ενημερωμένος και ποιοι όχι κύριε, και απευθύνουν στους ε, εκπροσώπους της Επιτροπής. Η κυρία Κλάστορ. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι το σκάνδαλο για το αλογίσιο κρέας δεν είχε να κάνει με την επισήμανση. Με την σήμανση. Ήταν μια απάτη, καθαρή απάτη. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω αυτά που είπε η Ρένα Ζόμερ. Δεν μπορούμε να πιστοποιούμε και αναφέρουμε όλο τον κύκλο ζωής του κρέατος. Γι' αυτό λοιπόν είμαι υπέρ της πρόθεσης της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω κατευθείαν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Φουστάγκεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι κι εγώ σύντομος. Αναφέρετε στο ψηφισμά σας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερεύει την εντολή της. Εγώ όπως τα φαντάζεστε, δεν συμφωνώ με αυτό και θα ήθελα να σας παραπέμψω στην αρχική νομική φάση 1069 του 2011, όπου γίνεται αναφορά στην κατάστασή μου για το βόλιο κρέας, αλλά ε, αναφέρεται και σαφήνεια ότι η ε, σήμανση προέλευσης μπορεί να διαφέρει από είδος κρέατος σε είδος κρέατος, ανάλογα με το ζώο και μπορεί αυτές οι διατάξεις, οι απαραίτητοι όροι να διαφέρουν α, ανάλογα το είδος κρέατος. Και θα πρέπει να λεφτεί υπόψη και τα τίτρα χαρακτηριστικά. Και ύστερα, στο 26.9, άρθρο 26.9 γίνεται αναφορά συγκεκριμένα σε μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά τον ε, τόπο εκτροφής και τον τόπο σφαγής. Με την νομική λοιπόν βάση αυτή, κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενέργησε μελέτη αντικτύπου και στο πλαίσιο αυτό είχαμε συνομιλίες και με τις εθνικές διοικήσεις και με τους εμπλεκομένους φορείς και προσπαθήσαμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία αφενός μεταξύ της ανάγκης ενημέρωσης των καταναλωτών για την προέλευση του κρέατος και αφετέρου του επιπρόσθετου κόστους, το οποίο συνεπάγεται προφανώς ε, μια τέτοια ρύθμιση για τον καταναλωτή. η μελέτη αντικτύπου που διενεργήθηκε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μεταξύ των διαφορετικών λύσεων η καλύτερη ισορροπία μεταξύ ε, κόστους και σκοπιμότητες ήταν να αναφέρεται το κάτω μέλος ως το κατάλληλο γεωγραφικό μοντέλο. Άρα, το να υπάρχει το μοντέλο του βόηου κρέατος, δηλαδή με τοπο γέννηση εκτροφής και σφαγής σε σύγκριση με ένα μοντέλο μόνο τόπου εκτροφής και τόπου σφαγής φαίνεται πιο περίπλοκο σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τους χείρους και τα εγωπρόβια. Ο κύκλος ζωής και παραγωγή είναι πολύ πιο σύντομος και τα υφιστάμενα συστήματα εντοπισμού δεν το επιτρέπουν αυτό σε όλες τις περιπτώσεις και σε ό,τι αφορά το διοικητικό άκτο το οποίο θα συνεπαγόταν, σε ό,τι αφορά τώρα τη σκοπιμότητα για τους καταναλωτές. Το εστιακό σημείο της ε, μελέτης ήταν ο τόπος εκτροφής. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα του Ευρωμαρομέτρου που θα δημοσιευθούν συντόμως που καταδεικνύουν ότι 88% των καταναλωτών στην Ευρώπη θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να είναι υποχρεωτικό ποσοστό αλλά μόνο ε, ένα μικρότερο ποσοστό θεωρεί ότι χρειάζεται και το πως Σε ό,τι αφορά αυτό το επιπλέον κόστο, εκτιμήθηκε ότι το επιπρόσθετο κόστος του να εφαρμοστεί το βόλιο μοντέλο θα ήταν 53% για το χείριο κρέας και 44% για, το ε, κρέας πτηνών και πουλερικών και αυτό θα συνεπαγόταν 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ επιπρόσθετο κόστος σε σχέση με, με το διπλό σύστημα, μόνο δηλαδή της χώρας εκτροφής και ε, σφαγής, που θα ήταν μόνο 800 εκατομμύρια. Δεν ε, χρειάζεται να διευκρινίσουμε ότι αυτό το κόστος τελικά μεταφέρεται και μετακυλείται στον τελικό καταναλωτή. Και τώρα μια τελευταία κουβέντα σε ό,τι αφορά ε, το μεταποιημένο κρέας, τον κοιμά ε, Το σχέδιο ψηφίσματος ε, αμφισβητεί και την αναφορά του τόπου προέλευσης μεταποιημένων τέτοιων προϊόντων. Αυτό θεωρούμε ότι δικαιολογείται από τη φύση των προϊόντων αυτών που συνδυάζουν διάφορες παρτίδες κρέατος. Αυτό γίνεται και είναι, υπάρχει ω δυνατότητα και στον ε, βόλιο τομέα. Σα δίνεται εντύπωση ότι αυτό δεν γίνεται στον τομέα του βόλου κρέατος, αλλά αυτό δεν ισχύει. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι παρέμεινε στο πλαίσιο της εντολής που της δόθηκε και ότι βρήκε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αφενός της ενημέρωσης του καταναλωτή και του ε, επιπρόσθετου κόστους και στο πλαίσιο αυτό η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των κρατών μελών και στο πλαίσιο των ε, διαδικασιών εφαρμογής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, έχει καταφτάσει και ο υπουργός. Θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα και θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια τον ε, Φεβρουάριο. Να καλωσορίσω τον Υπουργό, ο οποίος ε, έχει ήδη καταφτάσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα παρακαλούσα να καθίσετε στις θέσεις σας. Για να προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα ε, να καλωσορίσω εδώ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Τσαφτάρη. Θα ακολουθήσουμε την συνήθη διαδικασία. Θα γίνει μια παρουσίαση. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει ένας γύρος ερωτήσεων από πλευρά των συντονιστών και στη συνέχεια θα έχει την δυνατότητα ο Υπουργός να απαντήσει. Κατόπιν θα ξεκινήσει ένας γύρος ερωτήσεων για όλους τους συναδέλφους. Να παρακαλέσω εκ των προτέρων όλους τους συναδέλφους να είναι σύντομοι προκειμένου να έχουν όλοι οι συνάδελφοι τη δυνατότητα να πάρουν το λόγο και να απαντηθεί η ερώτηση τους. Σας ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Υπουργέ που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως. Έχουμε διάφορα θέματα εδώ στην Επιτροπή μας τα οποία τα συμπεριλαμβάνουμε στην ημερήσια διάταξη ασφαλώς οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί αλλά και σε ό,τι αφορά τους ε, σπόρους, σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία θα σας απασχολούν αναμφίβολα και εσάς και θα σας απασχολήσουν και στην Επιτροπή ε, Γεωργίας και στην Επιτροπή τη δική μας. Θα ήθελα όμως να δώσω σε εσάς την ευκαιρία να κάνετε την παρουσίασή σας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα με την ευκαιρία της ανάληψης της πέμπτης ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρουσιάσω στην Επιτροπή σας το πρόγραμμα στο πλαίσιο των εργασιών μας στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας η χρονική στιγμή που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερη και για τη χώρα μου και συμπίπτει με μια μεταβατική περίοδο για την Ευρώπη. Σε αυτό το σημείο καμπής το μεγάλο διακύβευμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζεται στην προώθηση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης ιδιαίτερα των νέων της Ευρώπης και στην εξασφάλιση σταθερότητας και ευημερίας για όλους τους πολίτες της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβεβαιώσει την αποστολή της και τη θέση της στην καρδιά και στη σκέψη των Ευρωπαίων πολιτών. Η προώθηση λοιπόν των πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη, την καταπολέμηση της ανεργίας, την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και των βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων η εμβάθυνση της ενοποίησης και η ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης καθώς και η αντιμετώπιση των εξωτερικών προκλήσεων όπως το μεταναστευτικό ζήτημα διαμορφώνουν το πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας. Οι θαλάσσιες πολιτικές της Ένωσης είναι μια θεματική που διατρέχει οριζόντια τις προτεραιότητές μας. Τώρα, ως, σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες στον τομέα της γεωργίας και της αλληλείας, γνωρίζετε όλοι μιλάμε για έναν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης, απασχόλησης, σε ό,τι αφορά τα, ε, τα θέματα της εξέτασης των εκθέσεων αυτών, πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι θα μπω στις λεπτομέρειες γι' αυτό, θέλω όμως να τονίσω ότι ο τομέας αυτός εξασφαλίζει την ποιότητα της διατροφής μας με σεβασμό στους φυσικούς πόρους που θέλουμε να τους διαχειριστούμε με αηφόρο τρόπο για να είναι το σύστημα βιώσιμο και φυσικά την προστασία του περιβάλλοντος όπως και την κοινωνία και το σεβασμό προς τους καταναλωτές έναν τομέα στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί την παγκόσμια διάκρισή της στις εξαγωγές με ισχυρούς κανόνες ασφάλειας, με αυστηρά πρότυπα παραγωγής που καταξιώνουν την εικόνα των ευρωπαϊκών προϊόντων. Αποφασίσαμε όλοι μαζί πρόσφατα τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής για να κάνουμε μεταξύ άλλων μια πράσινη, πιο πράσινη και πιο αποτελεσματική την γεωργία μας. Πρώτο μας μέλημα είναι λοιπόν η ολοκλήρωση αυτής της μεταρρύθμισης. Πρέπει να εγκριθούν έγκαιρα από την Επιτροπή η κατεξουσιοδότηση πράξης. Η Προεδρία ευελπιστεί ότι παρά τις αρχικές ανησυχίες η Επιτροπή θα καταλήξει σε κατεξουσιοδότηση πράξης που αντανακλούν πιστά την πολιτική μας συμφωνία σχετικά με τους νέους κανονισμούς της κοινή αγροτικής πολιτικής. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε δίνοντας τη δυνατότητα στους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν ομαλά την παραγωγική και επενδυτική τους προσπάθεια. Ταυτόχρονα πρέπει να, αξιολογήσουμε ορισμένα μέτρα της ΚΑΠ και να εντοπίσουμε τις αναγκαίες βελτιώσεις. Να ενισχύσουμε τη θέση των γεωργών και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην εμπορική διαδικασία, να τους φέρουμε πιο κοντά στον καταναλωτή προς αμοιβαίο όφελος ανφωτέρων. Στο Συμβούλιο σκοπεύουμε να εξετάσουμε την έκθεση που αναμένουμε από την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της αναθεώρησης του 2007 στον τομέα των φρούτων και λαχανικών και να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον του. Ο τομέας αυτός είναι σημαντικός όχι μόνο για την οικονομία και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για την υγιεινή διατροφή. Στο, στο ίδιο πλαίσιο η ελληνική προεδρία έχει στόχο να συζητήσει στο Συμβούλιο την έκθεση της Επιτροπής για το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα μετά τη λήξη των ποσοστώσεων. Ο φάκελος της προώθησης των αγροτικών προϊόντων είναι επίσης προτεραιότητα για την ελληνική προεδρία. Η εξέταση των προτάσεων που αναμένουμε από την Επιτροπή για την αναθεώρηση των μέτρων σχετικά με τα σχολικά προγράμματα διανομής γεωργικών προϊόντων στους μαθητές, την βιολογική γεωργία, όπως επίσης και τις προτάσεις για τις υπεραπομακρυσμένες μικρές νησιώτικες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του επόμενου εξαμήνου, όπως επίσης και η έκθεση για τη δημιουργία ενός προαιρετικού σήματος νησιωτικής γεωργίας σε σε ό,τι αφορά τώρα την έκθεση για την τοπική γεωργία και τις άμεσες πωλήσει που ήδη κατατέθηκε, αναμένουμε από την Επιτροπή να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα και να παρουσιάσει ενδεχόμενα νομοθετική πρόταση. Για την κοινή αλλιευτική πολιτική έχει ήδη επιτευχθεί πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και για τον κανονισμό της κοινή οργάνωσης αγοράς, με βασικό στόχο να εξασφαλίζεται περισσότερο βιώσιμη διαχείριση των πόρων. Για να ολοκληρωθεί όμως η μεταρρύθμιση, κύρια προτεραιότητά μας θα αποτελέσει η Συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Τα πολιτή σχέδια διαχείρισης, η Οργανωτική Ομάδα Εργασίας, η Task Force, οι εργασίες τις οποίες επιβεβαίωσαν την καλή θέληση και των δύο πλευρών και του Κοινοβουλίου αλλά και του Συμβουλίου να βρεθούν ρεαλιστικές λύσεις θα συνεχίσει τις εργασίες της με στόχο να έχουμε περαιτέρω αποτελέσματα ως το Μάρτιο του 2014. Μια άλλη προτεραιότητα αφορά στις εργασίες για την αφαρμογή της απαγόρευσης των απορρίψεων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής λάβαμε την πρόταση της Επιτροπής και σκοπεύουμε να προχωρήσουμε στην εξέτασή της. Η Προεδρία σκοπεύει επίσης να προωθήσει τις εργασίες για την τροποποίηση του κανονισμού για την αλληλευτική προσπάθεια στα βαθέα ύδατα, όπου και θα λεφτεί διόντως υπόψη το επικοδομητικό έργο το οποίο έχει ήδη αναλυφθεί από την πλευρά του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την υγεία των ζώων και των φυτών και την ασφάλεια γενικότερα της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Το Συμβούλιο δέχτηκε με ικανοποίηση από την Επιτροπή το πακέτο για ασφαλέστερα ζώα και φυτά και ασφαλέστερη αγροδιατροφική αλυσίδα που καλύπτει την υγεία των φυτών και των ζώων, το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, τους επίσημους ελέγχους στην αγροδιατροφική αλυσίδα και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πακέτο αυτό υιοθετήθηκε από την Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστούν πολύπλοκα θέματα στους επιμέρους τομείς αλλά και στην προσπάθεια για εξυγχρονισμό και απλούστευση του νομικού πλαισίου. Η συγκροτημένη και αποτελεσματική νομοθεσία έχει καθοριστική σημασία για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, την αξιοπιστία μεταξύ των εμπορικών εταίρων και φυσικά την βιωσιμότητα στην παραγωγή τροφίμων αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα ψηλότερα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων, οι κρίσεις που εμφανίζονται στην διατροφική αλυσίδα είτε πρόκειται για περιπτώσεις ανακριβούς επισήμανσης, είτε απάτης, είτε εμφάνισης ασθενειών των ζώων, μας αναγκάζουμε να προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας. Και οι πέντε προτάσεις του πακέτου έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και η ελληνική προεδρία θα δώσει υψηλή προτεραιότητα συνεχίζοντας το έργο των δύο προηγούμενων προεδριών του τρίου, τόσο της Ιρλανδικής όσο και της Λουθιανικής, λαμβάνοντας υπόψη και τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Η Ελληνική Προεδρία σκοπεύει να ολοκληρώσει την τεχνική έκθεση των επιμέρους προτάσεων και να συνταχθούν τα πρώτα συμβιβαστικά κείμενα τα οποία θα ενσωματώνουν τις απόψεις που εκφράζονται από τα κράτη-μέλη. Παράλληλα, η ελληνική Προεδρία σκοπεύει να παρακολουθεί στενά το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να διευκολύνει κατά το δυνατόν τις διοργανικές διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν επόμενη κοινοβουλευτική περιόδο. Ειδικότερα, ισότι ό,τι αφορά την πρόταση για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, η Ελληνική Προεδρία θα εργαστεί από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχειρώντας να ανοίξει το δρόμο για την επίτευξη μιας μελλοντικής συμφωνίας. Γνωρίζομαι πολύ καλά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από ορισμένους βουλευτές του Κοινοβουλίου αλλά και των πολιτικών ομάδων σχετικά με τις διάφορες προκλήσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση. Το Συμβούλιο εξετάζει προσεκτικά την πρόταση αναφορικά με τις επιπτώσεις και τις συνέπειές της. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για μια τέτοια πρόταση που έχει στόχο όπως τόνισα να εξυγχρονίσει και να απλουστεύσει ένα μεγάλο αριθμό λεπτομερών και τεχνικών μέτρων που ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια, απαιτείται αρκετή προσπάθεια ακόμη ώστε να πετύχουμε σαφείς κανόνες και νομική ασφάλεια, ακόμη και στη συνέχεια στο πλαίσιο των εξουσιοδιωτικών και των εκτελεστικών πράξεων. Τώρα, εις ό,τι αφορά την πρόταση για τον κανονισμό για την διαχείριση των δαπανών στον κτηνιατρικό και τον φυτο-υγειονομικό τομέα, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο εργάστηκαν σκληρά για να εξασφαλιστεί η έγκρισή της πριν το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου και για την επιτυχία της συμφωνίας σε πολιτικό επίπεδο. Η εξέταση της έκθεσης της Επιτροπής για την υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό σε τρόφιμα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά μας. Η Ελληνική Προεδρία είναι έτοιμη να αρχίσει άμεσα την εξέταση των προτάσεων σχετικά με την κλωνοποίηση των ζώων στο οποίο τον προ, τον στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου. Όλοι οι φορείς που έχουν ήδη εμπλακεί στη συζήτηση γνωρίζουν πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα. Η ελληνική προεδρία γνωρίζει επίσης την πρόσφατη συζήτηση στο ΚΟΜΕΜΒΗ σχετικά με την κλωνοποίηση των ζώων και θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Αναμένουμε ακόμη από την Επιτροπή της προτάσεις για τις οποίες η Ελληνική Προεδρία είναι έτοιμη να αρχίσει την τεχνική εξέταση εφόσον κατατεθούν σε εύκολο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές, τη δέσμη για την υγιεινή και την νομοθεσία για τα ζωοτεχνικά ζητήματα. Στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνονται θέματα ευθυγράμμισης με τη συνθήκη της Λισαβόνας, όπως του υφιστάμενου κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά. Αναμένεται σύντομα η πρόταση της Επιτροπής και η Προεδρία στοχεύει σε ένα επικοδομητικό διάλογο με την Επιτροπή τη δική σας για το θέμα αυτό. Τέλος, σχετικά με τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση και το δασικό τομέα, η προηγούμενη Προεδρία του Συμβουλίου ήδη συνέταξε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή κατευθύνσεων για την εφαρμογή της νέας δασικής στρατηγικής, η επεξεργασία του οποίου συνεχίζεται τώρα επί της και επί της ελληνικής προεδρίας. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, έκανα μια μικρή ανασκόπηση των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας σε μια σειρά από σοβαρά θέματα που έχουμε να χειριστούμε στους επόμενους μήνες στο πεδίο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλίας. Στη συγκυρία των ευρωεκλογών, μια ιερή και δηλωτική, όπως είπα, της δημοκρατίας διαδικασία που διέπει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί για μας πρόκληση να εργαστούμε με ρεαλισμό και με την πεποίθηση για ένα καλό αποτέλεσμα. Βασιζόμαστε για το σκοπό αυτό στη στενή συνεργασία, την ενεργό και αποτελεσματική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε, που είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους στόχους μας και από κοινού να βρούμε λύσεις για μια σειρά από σημαντικά και ευαίσθητε για την κοινωνία μας ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και κύριε Πρόεδρε με πολύ χαρά θα δεχτώ τις ερωτήσεις που ενδέχεται να έχετε εσείς ή και τα μέλη της Επιτροπής σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να διαβάσω ποιους ομιλητές έχω στον κατάλογο. Ροτ Μπέρεντ, ο συναδελφός Κουμουτσάκος, Κρίστα Κλάς, Δανέλης και Ζι Λέβενς. Ξέχασα κανέναν? Όχι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σειρά αυτή. Η κυρία Ροτ Μπέρεντ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω για δύο διαφορετικά ζητήματα τα οποία άπτονται των θεμάτων της Επιτροπής για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και για τα, τους κλόνους. Μία πρόταση έχουμε πριν από κάποια χρόνια ε, στις διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο απέτυχε η πρόθεση των θεμάτων αυτών γιατί τα κράτη-μέλη δεν ήταν διατέθημενα να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά ε, τα προϊόντα από κλωνοποιημένα ζώα. Μία πρώτη ερώτηση. Υπάρχει πλέον μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει, δεν περιλαμβάνει τίποτα, απολύτως τίποτα για την επισήμανση των προϊόντων των κλωνοποιημένων ζώων. Απαγορεύει μεν την εμπορία των κλωνοποιημένων ζώων, αλλά ποτέ δεν ήταν αυτό κανενός σκοπού. Ποτέ δεν θα ήθελε ένας παραγωγός να το κάνει αυτό, γιατί πολύ απλά κοστίζει πάρα πολύ. Μιλώντας για εμπορία, μιλάμε για δεύτερη και τρίτη γενιά προϊόντων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Αν η απαγόρευση δεν ε, επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την εμπορία στην διατροφική αλυσίδα. Συμφωνείτε μαζί, με, μαζί μου ότι τουλάχιστον θα πρέπει να επισημένονται τα προϊόντα που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα δεύτερης και τρίτης γενιάς για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, γνωρίζετε ότι είναι ακαθόδες το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπατε και εσείς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ψήφισε, υπερψήφισε ένα σχετικό ψήφισμα το οποίο σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι η έγκριση ενός γενετικώς τροποποιημένου καλαμποκιού του 1507 Pioneer δεν θα έχει συνέχεια. Θέλω να μου πείτε πώς ε, αντιμετωπίζετε αυτή την πρόταση αδειοδότησης. Θα το συζητήσετε τους επόμενους μήνες το θέμα αυτό και είσαστε διατεθειμένος να συζητήσετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουμε ενώπιόν μας. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα άλλο προϊόν έκρινε ότι δεν ε, ε, συμπεριφέρθηκε σωστά σε ό,τι αφορά την συμμετοχή σε ε, κράτη-μέλη και τις πατάτες Armflora. Και τώρα στα νέα προϊόντα επίσης έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη θέμα συμμετοχή των κρατών μελών, αλλά πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τι αμφιβολίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να δώσουμε τέτοια άδεια σε νέα προϊόντα, γιατί ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε απόλυτη βεβαιότητα. Και πολλοί κλάδοι ε, οικονομική και της ε, βιομηχανίας ε, το πιστεύουν αυτό και ένα προϊόν φοβόμαστε ότι ενδεχομένως να μπορέσει να προωθηθεί ένα προϊόν στις ΗΠΑ και μετά με τις εμπορικές συμφωνίες να εισαχθεί στις, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να το δούμε τον επόμενο χρόνο. Εγώ καλούμε να συνομοθέσω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να ξέρω αν συμφωνείτε για το συγκεκριμένο αραβόσιτο Pioneer 1507 ε, να μην δοθεί αδειοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ροτμπέρεντ ο συνάδελφος Κουμουτσάκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Ο τίτλος <clears throat> και η αρμοδιότητα της Επιτροπής <clears throat> προδικάζει σε μεγάλο βαθμό και την ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Και σχετίζεται και με ό,τι υπόθηκε <clears throat> προηγουμένως από την κυρία Συνάλφο σχετικά με τα κλωνοποιημένα ζώα και τα θέματα τα οποία προκύπτουν από αυτό το μεγάλο ζήτημα. Πρόκειται λοιπόν για την ασφάλεια τροφίμων και συγχρόνω την προάσπιση τη δημόσια υγεία. Γνωρίζετε βέβαια όπω και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες τα συγκλονιστικά γεγονότα τα οποία είδαν το φως τον τελευταίο καιρό σχετικά με τα σκάνδαλα στην ποιότητα τροφίμων. Διάφορα σκάνδαλα επαναλαμβανόμενα δημιουργούν ένα αίσθημα ανασφάλειας στον καταναλωτή και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αφορά τα ποιοτικά τρόφιμα, τα αγροτικά αλλά και τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Μαζί με αυτό αναδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό και η ανάγκη σωστής άρτιας πλήρους ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα και την προέλευση και την διατροφική αξία των τροφίμων. Είναι λοιπόν ένα θέμα κέρια σημασία για του Ευρωπαίου πολίτε και η ερώτησή μου είναι αν σκέφτεστε με την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προωθήσετε με κάποιο τρόπο, με κάποια συζήτηση, να πιέσετε πολιτικά για να υπάρχουν κάποια πιο συγκεκριμένα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση που αφορά, όπως είπα, το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών, ειδικά δε εν ώψη πολύ κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων των πιο κρίσιμων στην ιστορία της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ευρωπαϊκών εκλογών. Είναι ένα ζήτημα που καίει, καίει πραγματικά την, κοινωνία για τους Ευρωπαίους πολίτες η ποιότητα των, προφή, τροφίμων αλλά και το δικαίωμά τους να ενημερώνονται σωστά για την ποιότητα, για τη διατροφική αξία και για την προέλευση των προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κλάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, για την παρουσίαση του προγράμματός σας και σκέφτηκα ότι στις 18 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινά της ε, προεκλογική εκστρατεία και αυτό θα ε, περιορίσει σημαντικά το διάστημα συνεργασίας μας. Ε, ως Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θεωρώ ότι έχετε μια εγκάρσια τέτοια αρμοδιότητα η οποία άπτεται πολλών επιτροπών του Κοινοβουλίου. Καταρχάς για την κοινή αγροτική πολιτική. Σε αυτά θα ασχοληθεί ε, με αυτά θα ασχοληθεί η Επιτροπή ε, Γεωργίας και σε ό,τι αφορά τις ε, ε, πράξεις και σε ό,τι αφορά το πρασίνισμα, το greening αυτό. Εδώ ξέρετε οι απόψεις διήστανται και εγώ θα ήθελα να σας πω ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος ότι το πρασίνισμα δεν μπορεί να σημαίνει απλά πάυση κάθε δραστηριότητας. Θέλουμε ε, βιώσιμη εκμετάλλευση, βιώσιμη ανάπτυξη του πολιτισμικού τοπίου και αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτελεί στόχο της Προεδρίας. Θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα το οποίο δεν το θίξατε Μιλάμε για την αξιοποίηση των γεωργικών εκτάσεων, η γεωργία ως πηγή ενέργειας. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγεται μια συζήτηση για την... Ε, ολοκληρώθηκε μάλιστα σε πρώτη ανάγνωστη συζήτηση για τα βιοκαύσιμα και η Λιθωνική Προεδρία ε, δεν ε, κατάφερε να περάσει η πρόταση αυτή στο Συμβούλιο. Η ελληνική προεδρία, ακούγεται ότι θα το ξαναπιάσει το θέμα αυτό. Τι θα κάνετε λοιπόν, τι προγραμματίζετε να κάνετε, θα το ξαναπιάσετε το θέμα αυτό. Και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα βιοκαύσιμα. για τους παράγοντες ILOC θα κάνετε κάποιους, ε, κάποια πρόταση σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια και την ανάπτυξη βιομάζας. Αν θέλουμε να την προεκτήσουμε αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε να έχουμε και δική μας παραγωγή ενέργειας, χρειαζόμαστε ε, μια άλλη, ξέρετε, θεώρηση της ε, έμεσης αξιοποίησης των εκτάσεων. Τι προτίθεται λοιπόν να κάνει η Προεδρία από πλευρά της Ελλάδας ή το θέμα αυτό θα το αφήσουμε για την επόμενη Προεδρία μήπως. Μιλήσατε για το πολλαπλασιαστικό υλικό και εδώ βρισκόμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης και από πλευρά ε, τη Επιτροπή μα, αν και αρμόδια καθήλυνη η Επιτροπή ε, Γεωργίας. Δεν ξέρω τι πλεονεκτήματα υπάρχει από τη συνένωση 12 κανονισμών σε έναν. Και θα ήθελα να ξέρω όμως γιατί υπάρχει τόσο χρονική πίεση. Θα έπρεπε να έχουμε αρκετό χρόνο για τις διαβουλεύσεις. Ας πάρουμε το χρόνο που χρειαζόμαστε. Γιατί ξαφνικά είναι τόσο κατεπήγον αυτό το θέμα. Και προσπαθούμε τόσο γρήγορα να το πασαλείψουμε. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία για την Προεδρία σας που θα αποτελέσει επιτυχία και για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Δανέλης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θέλω να ευχηθώ στην Ελληνική Προεδρία να είναι επικοδομητική, αποτελεσματική και προωθητική στην αντιμετώπιση ε, πολλών από τα ζητήματα που απασχολούν το κοινό μας ευρωπαϊκό σπίτι. Ε, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι πολλοί εξημών θεωρούμε ότι η έκβαση της μεγάλης μεταρρύθμισης κοινή γεωργικής πολιτικής ως προς τον τομέα του πρασινίσματος ε, ήταν υποδέστερη των προσδοκιών και των φιλοδοξιών που στην αρχή της συζήτησης της μεγάλης μεταρρύθμισης είχαμε. Σχετικά λοιπόν με αυτή την πραγματικότητα και γνωρίζοντας τις δικές σας προσωπικές ευαισθησίες στα ζητήματα αυτά, πώς βλέπετε η ελληνική προεδρία μέσω της ε, πρόθεσης των εφαρμοστικών πράξεων που έχετε μπροστά σα. Και είναι μια μεγάλη πρόκληση και μια μεγάλη ανάγκη να επισπευστεί και να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια τη Προεδρία. Πώ βλέπετε να υποστηρίζετε και να αξιοποιείτε στο έπακρο η δυνατότητα παροχή δημοσίων αγαθών που έχουν σχέση ε, με την αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή και την προάσπιση του περιβάλλοντο και πιο συγκεκριμένα πώς βλέπετε την αξιοποίηση του εργαλείου ε, που θεωρώ ότι είναι καθοριστικό στην αλλαγή αντίληψης πρακτικών ε, στην γεωργία, την αξιοποίηση του εργαλείου των ε, μηχανισμών υποστήριξης των αγροτών και κυρίως των νέων, της μετάβασης, της μεταφοράς της γνώσης, της καινοτομίας, της εξυπηρέτησης στο επίπεδο της παροχής των υπηρεσιών γνώσης που τόσο λείπει από, από πολλές από τις χώρες μας και βεβαίως ε, χαρακτηρίζει κυρίως τους, ε, τον αγροτικό πληθυσμό μιας περασμένης ηλικία και τη μεγάλη αναγκαιότητα της μετάβασης σε ένα άλλο, ε, σε ένα άλλο προσωπικό άσκησης της γεωργίας. Ευχαριστώ πολύ. Vielen Dank, Um, Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για μια πλήρη παρουσίαση. Ένα από τα μηνύματά σας είναι ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά με τους καταναλωτές και γνωρίζω ότι τους τελευταίους μήνες τα θέματα τα μεγαλύτερα στα οποία και οι εκλογείς μου ενδιαφέρονται αφορά καταρχάς το θέμα της ποράς και φυσικά τα γενετικά τροποποιημένα. Ιδιαίτερα το θέμα των γενετικά τροποποιημένων θα με απασχολήσει. Την προηγούμενη Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, υπερψήφισε και με μεγάλη πλειοψηφία την πρόταση που έκανε η πολιτική μου ομάδα που απέριπτε την πρόταση αδειοδότησης γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού. Ένας από τους λόγους είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπέρασε τις εφαρμοστικές της δυνατότητες και στην περίπτωση της ανφλόρα, της πατάτας και στην περίπτωση του καλαμποκιού. Οι διαδικασίες δεν έγιναν σεβαστές γιατί μετά από την τροποποίηση της πρότασης αδειοδότησης δεν διαβουλεύτηκε με την αρμόδια επιτροπή. Είναι σαφές λοιπόν ότι αυτή στιγμή έχει αλλάξει η ε, πρόταση από την αρμόδια επιτροπή και την απόφασή της, τότε θα πρέπει να επανέλθει το θέμα προς εξέταση κάθε φορά και η πρόταση. Το θέμα είναι ότι η Προεδρία έχει θέσει το θέμα αυτό σαν βασικό θέμα στο επόμενο ΕΚΟΦΗΝ θα ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλει την τροποποιημένη πρόταση στην αρμόδια Επιτροπή για ψηφοφορία έτσι ώστε να αποφύγετε στο μέλλον νομικού τύπου αμφισβητήσεις. Το θέμα αυτό πρέπει να απασχολήσει και το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν συζήτηση και ζητάμε από την Ελλάδα που έχει μια σκληρή θέση σε σχέση με μια γεωργία ελεύθερη γενετικά τροποποιημένων να προχωρήσει στο θέμα. Σε ευχαριστώ. Πίλαρ. Φλόρεντς. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που μας εξηγήσατε το πρόγραμμά σας, ένα πρόγραμμα πάρα πολύ πυκνό και θα ήθελα να σας ευχηθώ μια εξαιρετική προεδρία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς είστε και υπουργό και για θέματα γεωργίας και για θέματα τροφιμικής ασφάλειας. Και ίσως να έχετε μια συνολική ιδέα θα έλεγα, την οποία θα χαρακτήριζα οριζόντια των προβλημάτων που μας απασχολούν πρέπει να, απασχολήσουμε, να, ε, να διαπιστώσουμε ότι η ασφάλεια στα τρόφιμα είναι εξαιρετική στην Ευρώπη. Έχουμε νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά πλήρεις, μπορώ να πω ότι είναι οι καλύτερες στον κόσμο, έτσι ώστε να αποτρέψουμε πιθανά προβλήματα μέσω ε, της, ε, της διατροφής. Βέβαια αυτό δεν αποκλείει τις απάτες οι οποίες μπορεί να γίνουν. Και θα ήθελα να θέσω κάποια επιπλέον θέματα. Στο θέμα της ασφάλειας των τροφίμων, εμείς είμαστε αυστηροί όπως είπα στην νομοθεσία μας και υπάρχουν πάρα πολλοί γεωργοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί σε χώρες όπως η δική μου, χώρες του Νότου, ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλά έντομα εν πάση περιπτώσει, και η νομοθεσία για τα εντομοκτώνα, έτσι όπως προβλέπετε. Ε, δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια προϊόντα τα οποία θα μας ήταν χρήσιμα για να καταπολεμήσουμε τη μάστιγα των εντόμων. Και αυτό επηρεάζει αρνητικά τους γεωργούς. Είναι ένα από τα πολλά προβλήματα τα οποία έχουμε και αυτό προκαλεί υπερβολικό κόστος για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Σχετικά τώρα με τις ετικέτες προέλευσης ε, του κρέατος, όταν το κρέας χρησιμοποιείται σαν ένα επιπλέον συστατικό. Θα ήθελα και τις απόψεις σας για αυτό το θέμα. Μια νομοθεσία η οποία θα πρέπει να απαιτεί την ετικετοθεσία κρέατος ως συστατικού, σαν παράδειγμα και το κρέας αλόγου είναι ένας κανόνας ο οποίος δεν ξέρω πώς μπορεί να εφαρμοστεί γιατί είναι ιδιαίτερος περίπλοκος. Και αυτά τα είχαμε πει και με την κυρία Τεστόρη της ΣΑΝΚΟ. Και αναφέρομαι στη χρήση του κρέατος σε μεταποιημένα προϊόντα, σε προϊόντα επεξεργασμένα. Τώρα, υπάρχει άλλο ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο και το οποίο θα περάσει και στην επόμενη νομοθετική περίοδο γιατί αναμειγνύεται και με άλλα θέματα όπως τα γενετικά τροποποιημένα, η συζήτηση η οποία γίνεται επίσης για την οικολογική γεωργία, η απλούστευση της νομοθεσίας και επίσης και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερως οι μικρή παραγωγή. Θα ήθελα την άποψή σας λοιπόν για τους μικρούς παραγωγούς. Να καθορίσουμε σωστά τι είναι ένας μικρός παραγωγός, ο οποίος ε, εμπορεύεται τοπικές παραδοσιακές ποικιλίε και ποια είναι και η αγορά των σπόρων που συνδέεται με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν ε, φυσικά πάρα πολλές μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες για τη σπορά που παράγουν σπόρους αλλά υπάρχουν επίσης και πάρα πολύ μικρές τέτοιες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις επιμέρους παραγωγές. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει εμείς ε, να έχουμε μια νομοθεσία που να καλύπτει τις ανάγκες και των μεν και των δε. Γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουμε μια παράλληλη αγορά εκτός κάθε ελέγχου Πρέπει λοιπόν εμείς να βοηθήσουμε στον τομέα της σποράς και τους μικρούς παραγωγούς έτσι ώστε να αποτρέψουμε τη δημιουργία μιας παράλληλης ανεξέλεγκτης αγοράς. Ο συνάδελφος Καλ Χάιντς Φλόρεντς, κύριε Υπουργέ, με ακούτε? Ωραία. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για την Προεδρία. Θα ήθελα να τονίσω ότι ως Γερμανός χαίρομαι ιδιαιτέρως που αναλάβετε την Προεδρία. Δεν είναι απλά τα πράγματα, το γνωρίζουμε. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας υποστηρίξουμε. Μία ερώτηση έχω να κάνω, η οποία είναι πάρα πολύ ε, βαρετή. Την θέτω εδώ και 20 χρόνια σε όλους τους υπουργού. Έχουμε μία τεράστια συμφωνία εδώ στο Κοινοβούλιο για πάρα πολλά θέματα, για πολλά έχουμε αποφασίσει, αλλά πάρα πολλά δεν εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε καμία ιδέα πώς αυτά που αποφασίζουμε εδώ από κοινού μπορούν επιτέλους να εφαρμοστούν. Γιατί δεν χρειάζεται να έχουμε τα κορυφαία πρότυπα πάντα σε όλα τα θέματα, αλλά να έχουμε ενιαία πρότυπα. Ξέρετε λοιπόν, υπάρχουν ε, στη Γερμανία, στην ε, Βέλγιο, στην Ολλανδία, ε, υπάρχει διαφορά ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των, πρωτο, των προτύπων. Και αν ρωτιόμαστε λοιπόν, έχετε λοιπόν μια ιδέα για το πώς γίνονται τα πράγματα. Σας ευχαριστώ και τελευταίος ε, και παρακαλώ την συντομία ο συνάδελφος Χρυσόγελος. Ναι κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι είναι επίκαιρα μερικά θέματα τα οποία έχουν δείξει και άλλοι συνάδελφοι. Ε, το θέμα με το Καλαμπόκι 1507 που πρέπει να διαχειριστείτε εσεί πολύ σύντομα και δεν πρέπει στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας να ανοίξει πόρτα για καλλιέργεια γενετικά τροπημένου καλαμπόκιου μετά από πολλά χρόνια διαδικασίας. Ε, είστε ενήμερος για αυτό το θέμα από τον ε, Δεκέμβριο. Νομίζω και εγώ σας είχα θέσει αυτά τα θέματα. Υπάρχει το θέμα με το μέλι, με την οδηγία για το μέλι. Ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ τους μελισσοκόμους ε, και τους καταναλωτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια το Κοινοβούλιο ψήφισε εκείνη τη διάταξη που αναγράφεται η παρουσία γυρισε από τροποποιημένα είδη όταν είναι συγκέντρωση από 0,9% και πάνω. Ε, Παρ' όλα αυτά εσείς ως ε, Συμβούλιο πρέπει να συζητήσετε αυτά τα θέματα και να μας δώσετε μία απάντηση. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο αναμένεται και στα πλαίσια του διαλόγου με τις ΗΠΑ να απασχολεί στο Συμβούλιο και θα θέλαμε τη γνώμη του Συμβουλίου και, του Προεδρία και της Προεδρίας του Συμβουλίου αφορά τα κλωνοποιημένα ζώα και τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τα κλωνοποιημένα ζώα αλλά και του απογόνους κλωνοποιημένων ζώων. Εάν έχετε επεξεργαστεί κάποια στρατηγική για το θέμα, ξέρουμε καλά ότι υπάρχει μεγάλη πίεση από τις ΗΠΑ στην Κομισιόν να μην αναγράφεται η προέλευση ε, να μην αναγράφει δηλαδή ότι τα, τα προϊόντα προέρχονται από κλωνοποιημένα ή από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν έχει γίνει μια προετοιμασία. Και τέλος, ε, εάν έχει γίνει προετοιμασία και παρακολούθηση εφαρμογή απαγόρευσης για δύο χρόνια της χρήσης των νέων, νοικοτινοειδών ε, φαρμάκων τα οποία ξέρουμε ότι βλάπτουν και τις μέλισσες. Έχει γίνει πολλή συζήτηση εδώ και σε αυτήν την Επιτροπή εάν έχετε παρακολουθήσει τη διαδικασία ως Συμβούλιο, αν τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ε, την απαγόρευση, αν έχετε στοιχεία για όλα αυτά, ε, να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο Υπουργό θα έχει τον λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και πάλι και ευχαριστώ όλους για τις πολύ χρήσιμες συζητήσεις, για τις ερωτήσεις θα αρχίσω από τις τα γενικότερα θέματα που θίχτηκαν, όπως αυτά που αφορούν τη γενικότερη παραγωγική διαδικασία και της, της Ευρώπης, την νέα κοινή αγροτική πολιτική και τα επιμέρους της θέματα και θα πάω σε πιο εξειδικευμένα θέματα όπως αυτά των κλωνοποιημένων ζώων, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, του μελιού κλπ. Αρχίζω από το γενικότερο που αναφερθήκατε κι εσείς κύριε Κουμουτσάκου. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη, ακόμη ακόμα και η δική μου η μικρή χώρα η Ελλάδα, έχει ένα ποικιλόμορφο περιβάλλον και παράγει ποικιλία πολλών ποικίλων εξαιρετικής ποιότητος προϊόντων. Μπορούμε να μιλούμε για την ελληνική γεωργία αλλά είναι διαφορετική η ελληνική γεωργία σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου από ότι είναι η ελληνική γεωργία στα βουνά της Υπήρου και από ότι είναι η ελληνική γεωργία στον κάμπο της Θεσσαλίας. Το ίδιο, το ίδιο πρότυπο αν το μεγέθυνα θα ίσχυε για όλη την Ευρώπη. Η ποικιλομορφία των αγροτικών συστημάτων της Ευρώπης είναι το ιδίωμά της, είναι το ιδιαίτερο πλεονέκτημά της και μάλιστα η Ευρώπη έχει πολιτικές που θέλουν να υποστηρίξουν αυτήν την παραγωγική διαδικασία και τα σήματα ποιότητας. Δεν είναι τυχαίο που η Ευρώπη καθιέρωσε για να υποστηρίξει αυτά τα συστήματα τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης, το σήμα με τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, το σήμα με τα προϊόντα του βιολογικού τρόπου παραγωγής, ενώ έρχονται ακόμα τρία τέτοια σήματα όπως αυτά της νησιώτικης παραγωγής που αναφέρθηκα και στην εισαγωγή μου, όπως αυτά της ορεινής παραγωγής και το σήμα με τα παραδοσιακά προϊόντα της Ευρώπης που δείχνουν την πολιτική της να υποστηρίξει αυτή την ποιότητα με μέτρα και, ε, και θεσμούς. Μάλιστα και εμείς δουλεύοντας προς το σκοπό αυτό αποφασίσαμε στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών που θα λάβει χώρα στην Αθήνα στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας μεταξύ της 4ης και 6ης Μαΐου αυτό να είναι το θέμα συζήτησής μας. Να δούμε πώς αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα της ποικιλομορφία των συστημάτων παραγωγής που αντανακλάται στην ποικιλομορφία των προϊόντων της Ευρώπης θα, γίνει, θα μετατραπεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα της Ευρώπης έναντι των ανταγωνιστών της. Σε ό,τι αφορά το θέμα της κοινή αγροτικής πολιτικής που έθιξε και ο κύριος Δανέλης. Νομίζω ότι τα κοινά χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικής που συναποφασίσαμε άλλωστε όλοι μαζί δείχνει για πρώτη φορά ότι θα δοθούν, θα εξακολουθήσουν να δίδονται σημαντικοί πόροι της Ευρώπης για να υποστηριχθεί η γεωργία σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο της συμφωνίας. Να υποστηριχθεί η παραγωγή αυτή καθεαυτή. Να υποστηριχθεί το πρασίνισμά της. Και θα έρθω ιδιαίτερα σε αυτό γιατί θύχτηκε και από την κυρία Κλάς. Να υποστηριχθούν οι νέοι αγρότες. Να μην αγνοούμε ότι η δημογραφική γύρανση του αγροτικού πληθυσμού επηρεάζει οριζόντια σχεδόν το σύνολο της ευρωπαϊκής παραγωγής και δεν είναι τυχαίο που ομόφωνα είπαμε ότι μέχρι και 2% των χρημάτων από τη νέα ΚΑΠ θα πρέπει να δοθούν για να υποστηριχθεί η είσοδος νέων ανθρώπων στην αγροτική παραγωγική διαδικασία γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε μπορεί να τα καταφέρουμε στη γεωργία με λιγότερο ίσως νερό, με λιγότερο ίσως και ακριβότερη ενέργεια ή κάποιο λίπασμα. Δεν μπορεί να υπάρξει όμως γεωργία χωρίς αγρότες. Γι' αυτό και θα πρέπει να δώσουμε και δίνουμε επισταμένη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή κύριε Δανέλη. Εις ό,τι αφορά τις άλλες προκλήσεις που έβαλε μπροστά μας η κοινωνία και αντιμετωπίζονται με την, στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ. Να αντιμετωπίσουμε πιο προσεκτικά τις ανάγκες, να ακούσουμε πιο καλά τις ανάγκες των καταναλωτών, μπορούμε να προλάβουμε την εκδήλωση προβλημάτων μέσω σωστότερης διατροφής και επίσης να ετοιμαστούμε, αυτό είναι και η μεγάλη πολιτική μπροστά στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2.20 για την Ευρώπη, να ετοιμαστούμε για, την, για τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές, όχι μόνο να τις απαλύνουμε όσο μπορούμε να τις περιορίσουμε, αλλά και να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Και η χώρα μου, μιλώντας τώρα με την ιδιότητα του Έλληνα Υπουργού Γεωργίας, είναι η πρώτη που νιώθει ήδη στο πετσί της, στο σώμα της, τις επερχόμενες αυτές κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις της στη γεωργία. Θα δείτε την ακαρπία των δέντρων ένα εκατονίπιων χειμώνων που αρχίζουμε να έχουμε στη χώρα μας. Βλέπουμε νέα είδη, νέα νέα έντομα, νέες αρρώστιες να έρχονται από πιο νότια κλπ. Σίγουρα ο μόνος τρόπος να κάνουμε βιώσιμα τα μελλοντικά αυτά σχήματα είναι μέσω της επιστήμης, της γνώσης, της έρευνας, της τεχνολογίας, της αξιοποίησης του τόπιου πλούτου, της βιοποικιλότητας που έχουμε. Έχουμε γενετικό υλικό και με αυτό θα ήθελα να τονίσω ξανά τη σημασία αυτής της βιοπικιλότητας. Είναι πλούτος που μπορεί να αξιοποιηθεί αύριο καλύτερα. Επομένως θα αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία είτε αφορά την έρευνα και τη γνώση, την εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα το εργαλείο των συμβούλων που πρέπει να έχει δίπλα του ο αγρότης έτσι ώστε γρήγορα να, να περάσει αυτή η γνώση προς τον αγρότη, όπως επίσης και το νέο εργαλείο που αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι οι λεγόμενες συμπράξεις καινοτομίας το clustering όλων των stakeholders σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, από τις εισρωές, από τον αγρότη, από τον μεταποιητή, τον διακινητή μέχρι τον καταναλωτή, προκειμένου γρήγορα μέσω αυτού του εργαλείου να ενσωματώνεται νέα γνώση και καινοτομία στον παραγωγικό τομέα. Και σε ό,τι αφορά το ειδικότερο θέμα που θύχτηκε για την ΚΑΠ και αφορούσε το πρασίνισμα. Η, απέτηση της νέας ΚΑΠ να ξοδευτεί έστω 30% των πόρων με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθούνται φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές ήταν μια σημαντική πολιτική απόφαση και σηματοδοτεί ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στείνουν ο νους και ακούν τα μηνύματα της κοινωνίας και ιδιαίτερα των μελλοντικών γενεών γιατί η αηφορία αυτό σημαίνει πρέπει να ακούσουμε αυτά που θα πούν οι μελλοντικέ γενιές. Και αυτές λένε πρέπει να έχουμε και εμείς νερό, να έχουμε και εμείς έδαφος καθαρό, να παράξουμε και εμείς. Επομένως, οι πρακτικές που βάζει μέσα ήδη στις αποφάσεις της η κοινή αγροτική πολιτική δηλώνουν τους τρόπους που επιθυμεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Για παράδειγμα, λέει να, να, να γίνει εναλλαγή των καλλιεργειών να αποφεύγουμε στο ίδιο έδαφος να καλλιεργούμε μονίμως τις ίδιες καλλιέργειες. Όλοι γνωρίζουμε ότι η αναλλαγή καλλιεργειών είναι πιο αηφόρα από την συνεχή μονοκαλλιέργεια. Να βάλουμε πολιετής καλλιέργειες. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πολιετής καλλιέργεια είναι προτιμότερη από την μονοητή γιατί μια φορά οργώνεις ένα χωράφι που θα μπει τριφύλι και για δέκα χρόνια δεν θα το ξαναοργώσεις η καλλιέργεια των ψυχανθών που δίδεται ιδιαίτερη έμφαση και δίδει τη δυνατότητα να αυξηθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις 2% επιπλέον εφόσον στο χωράφι μπαίνει ψυχανθές φυτό. Για τρεις λόγους. Όχι μόνο να εξασφαλιστεί ντόπια ευρωπαϊκή ζωοτροφή, πρωτεϊνούχος ζωοτροφή στην Ευρώπη για την κτηνοτροφία της, όχι μόνο να εξασφαλιστεί τροφή με όσπρια στο τραπέζι της ευρωπαϊκής διατροφής, ένα σημαντικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής που όλοι τώρα υποστηρίζουμε, αλλά και για περιβαντολογικούς λόγους. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μειώσεις το κόστος παραγωγής, να μειώσεις την εισρωή, την, το, το κόστος λιπασμάτων, να μειώσεις τη χρήση ε, χημικών λιπασμάτων από το να καλλιεργήσεις ψυχανθή, γιατί αυτά παίρνουν μόνα τους το άζωτο από την ατμόσφαιρα. Να λοιπόν οι τρόποι που μπορούμε υλοποιώντας τους να πάμε σε πιο πράσινες πολιτικές. Σε ό,τι αφορά τα, τα, θέματα που θύχτηκαν για, τα, για την βιολογική γεωργία, για τα θέματα με τις μικρές επιχειρήσεις και τους παραγωγούς, σας είπα ότι μέσα στην κοινή αγροτική πολιτική ένας τρόπος να τους βοηθήσεις αυτούς τους ανθρώπους πρώτον είναι να απλουστέψεις τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και στην κοινή, στη νέα ΚΑΠ προβλέπονται διεργασίες όπου κάτω από ένα ορισμένο μέγεθος της εκμετάλλευσης κάτω από ένα πόσο χρηματοδότησης σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις. Δεν χρειάζονται γραφειοκρατικές διεργασίες για τους μικρούς και αυτός είναι ένας τρόπος βοήθειάς τους. Η καθιέρωση των farmers market, των short supply chains, των κοντών της, της μικρής αλυσίδας αγοράς όπου φέρνουν εύκολα την παραγωγή μιας μικρής εκμετάλλευσης κατευθείαν στην, ε, στην κατανάλωση. Είναι εργαλεία που δουλεύουν προς την κατεύθυνση που κι εσείς επισημένατε, Δηλαδή να υποστηριχθεί και η μικρή γεωργία που ήταν παράδοση και είναι και ακόμα κομμάτι της ραχοκοκαλιάς της ευρωπαϊκής γεωργίας. Σε ό,τι αφορά τις πολυπλοκότητες ε, που θύχτηκαν και τις, ε, ε, πάλι με τον, για το σχετικό θέμα και από τον Γερμανό Ευρωβουλευτή επαναλαμβάνω, κάτι θα είναι εφαρμόσιμο όσο είναι απλούστερο. Όσο απλούστερο είναι, τόσο πιο εύκολα μπορεί και ο μικρός να το εφαρμόσει. Αλλιώς όταν γίνεται πολυπλοκότερο, μπορεί να το εφαρμόσει ο μεγάλος, αλλά είναι δύσκολα να το εφαρμόσει ο μικρός. Και τέλος, για το συγκεκριμένο θέμα, θέλω να θίξω ότι πάντοτε όταν φτιάχνουμε οριζόντιες ρυθμίσεις, υπάρχουν καταστάσεις που κάποιο κράτος έχει ιδιαιτερότητες και δυσκολίες να τον εφαρμόσει. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που μας απασχολεί και αφορά τις εκφορτώσεις στα πλαίσια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Είναι εύκολο ένα κράτος να ψαρεύει μόνο ένα μεγάλο είδος, ας το πούμε μπακαλιάρο, είναι εύκολο να το εκφορτώσει αυτό και να το ελέγξει μόνο σε ένα λιμάνι. Επομένως μια χώρα που ασκεί αυτή την αλλιευτική διεργασία είναι εύκολο να τον εφαρμόσει. Στη χώρα μου όμως που αλλιεύουμε 30 ή περισσότερα διαφορετικά είδη σε μικρές ποσότητες και θα κληθούμε γιατί τα εκφορτώνουμε σε 150 λιμάνια, δέστε τι δυσκολίες θα έχει η εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Άρα και εκεί θα πρέπει να ισχύσει η αρχή των ορίων. Δεν έχει νόημα να ψάχνουμε να ξοδεύουμε 100 ευρώ για να δούμε μισό κιλό ενός ψαριού που το κόστος του θα είναι πολλαπλάσιο για να το μετρήσουμε και να εφαρμόσουμε το συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πιο εξειδικευμένα θέματα που θύχθηκαν, αυτά της κλωνοποίησης που όπως υπόθηκε απασχολούν όλους, έχω ήδη αναφερθεί, η συζήτηση για τις προτάσεις αυτές Άλλωστε όπως γνωρίζετε μόλις κατετέθησαν την 19η Δεκεμβρίου ήρθαν από την Επιτροπή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα στο πλαίσιο του Συμβουλίου και των προκατε... προπαρασκευαστικών οργάνων του. Όμως θα ξεκινήσουν άμεσα. Δεν υπάρχουν επομένως πολλά που μπορούμε να πούμε σε αυτό το στάδιο για το περιεχόμενό του σαν Συμβούλιο. Η Προεδρία σκοπεύει, όπως είπα, να ξεκινήσει την εξέτασή του στα όργανα του Συμβολίου άμεσα και έχουν ήδη προγραμματιστεί οι συγκεκριμένες ημερομηνίες. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, που ε, και αυτό θύχτηκε και είναι ένα σημαντικό θέμα και απασχολεί και την κοινωνία μας. Όπως γνωρίζετε καλά, από το 2010 άλλωστε αναφέρθηκε ήδη, δεν έχει εγκριθεί καμιά γενετικά τροποποιημένη ποικιλία φυτών για καλλιέργεια. Ακόμα και η τελευταία που ήταν η πατάτα αμφλόρα που κι εσείς αναφέρετε, της οποίας η έγκριση ακυρώθηκε από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Δεκεμβρίου του 2013, δηλαδή πρόσφατα. Επομένως, η μόνη εγκεκριμένη καλλιέργεια παραμένει το καλαμπόκι της Μονσάντο, το γνωστό Μονσάντο 810, της σε εκκρεμεί μάλιστα η ανανέωση της έγκρισης εδώ και αρκετά χρόνια. Γνωρίζετε ότι, το, τη θέση των καταναλωτών. Ίσως ό,τι αφορά το καλαμπόκι 1507 που, που είναι επίσης μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση που θύχτηκε, αφότου το σχέδιο της απόφασης κατατέθηκε από την Επιτροπή μετά τη γνωστή δικαστική απόφαση που αναφερθήκατε, και απασχολεί πλέον την Προεδρία μας, ακολουθήσαμε τη γνωστή διαδικασία με την εξέταση στο Κορεπέρ. Σήμερα εξετάζεται σε τεχνικό επίπεδο και την Παρασκευή σε επίπεδο Κορεφέρ πάλι θα δηλωθεί θέλουμε να δούμε την πρόθεση ψήφου των κρατών μελών. Η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη, καθορίζεται από τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Συμβουλίου και όπως ξέρετε η Προεδρία δεν έχει καμιά δυνατότητα να παρεκκλίνει από αυτούς τους κανόνες και θα το σεβαστούμε απόλυτα. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον θέμα των, ε, του μεγάλου πακέτου για τα ασφαλέστερα ζώα και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη αν παίρνω ένα λεπτό παραπάνω αλλά υπήρξε πληθώρα ερωτήσεων και προσπαθώ να απαντήσω όσο το δυνατόν περισσότερες για το μεγάλο πακέτο για τα ασφαλέστερα ζώα, τα φυτά κλπ. Ειδικά για το θέμα που αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό, το αναπαραγωγικό υλικό, η Ελληνική Προεδρία, όπως είπα, θα εργαστεί από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ανοίξει το δρόμο για την επίτευξη μιας μελλοντική συμφωνίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από ορισμένου βουλευτές του Κοινοβουλίου αλλά και των πολιτικών ομάδων σχετικά με τις διάφορες προκλήσεις που προτείνονται στην πρόταση. Το Συμβούλιο την εξετάζει προσεκτικά αναφορικά με τις επιπτώσεις και τις συνέπειές της. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι σημαντικές για μια τέτοια πρόταση όπως και εσείς επισημάνατε Επι οποία όμως έχει στόχο να το εξυγχρονίσει και να απλουστεύσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό λεπτομερών και τεχνικών μέτρων που ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια απαιτείται αρκετή δουλειά, συμφωνώ μαζί σας, ώστε να επιτύχουμε σαφείς κανόνες και νομική ασφάλεια, συμπεραλαμβανομένων και εκείνων που θα καθοριστούν στη συνέχεια με εξουσιδιωτικές και εκτελεστικές πράξεις. Για την ελληνική προεδρία όμως αποτελεί ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο θα εξεταστεί διεξοδικά αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τον όποιο χρόνο διαθέτουμε στη διάρκεια της Προεδρίας μας. Και θα δουλέψουμε σκληρά γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να πάρω περισσότερο χρόνο κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Θα έχουμε και την ευκαιρία για τους διαφόρους φακέλους να ξανασυζητήσουμε τους επόμενους μήνες από πλευράς από τις Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έχουμε πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί αν δεν το καταφέρουμε δεν θα υπάρχει συνέχεια την οποία επιθυμούμε να υπάρχει και θα πρέπει να ξαναξεκινήσει η δουλειά από την αρχή στην επόμενη θητεία. Σας εύχομαι και σε σας καλή επιτυχία για τους επόμενους μήνες. Ε, πολύ δύναμη, επιμονή και υπομονή γιατί είναι μαραθώνιος ο δρόμος. Είναι ε, ξέρετε και πιο περιορισμένο ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή σα για να καλύψετε την ίδια απόσταση. Μέχρι τον Απρίλιο έχουμε και μετά ξεκινάει η προεκλογική διαδικασία για μα και σα εύχομαι συνολικά κάθε επιτυχία για την Προεδρία. σα το είπα και στον Υπουργό Υγεία πριν από λίγο. Χαίρομαι ιδιαίτερω που η Ελλάδα ανέλαβε την Ευρωπαϊκή Προεδρία και χαίρομαι που τα πράγματα οδεύουν ανωδικά. Και πάλι ξέρουμε ότι πολλά ε, χρειάστηκε να γίνουν για να εξέλθουμε από την κρίση και θα ήθελα και να σας πω ότι συμπαθώ προσωπικά και την Ελλάδα, όχι μόνο επειδή κάνω διακοπές, αλλά πρόκειται και για την πιο ε, παλαιά δημοκρατία και λοιπόν σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.